Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε στο σεμινάριο αυτό όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση των ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ και ελπίζουμε να βρείτε το σεμινάριο αυτό ενδιαφέρον και την ε, ανταλλαγή απόψεων που θα έχετε με τους ευρωβουλευτές και με όλους τους άλλους φορείς και παράγοντες που ασχολούνται με το θέμα. Ό,τι βρείτε λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για το πρόγραμμά μας, για τα σεμινάρια κλπ. Οι δύο συνάδελφοι που είναι εδώ δεξιά μου, Παύλα Φερνάντη Σέρβας, είναι και υπεύθυνη για την οργάνωση των ε, σεμιναρίων. Είναι από την Ισπανία. Εγώ είμαι Έλληνας. Έχουμε και από την Βουλγαρία τον Ντότσο Κολάκοφ που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Για μια ομάδα ε, βοηθών στην υπηρεσία μου που συνέφεραν και αυτοί. Δεν είναι εδώ στην αίθουσα αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα θα σας δοθεί ευκαιρία. Να, η Βάλτα είναι εκεί με το κίτρινο. Η κυρία με το κίτρινο. Η Μαρλίν Λέμενς κάθεται επίση εκεί, ντυμένη στα μπλε, που βοήθησαν και βοηθάνε γενικά την οργάνωση τέτοιων σεμιναρίων και είναι στη διάθεσή σας για ό,τι οι απορίες ή προβλήματα μπορεί να έχετε σχετικά με την οργάνωση. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη πρόγραμμα οργάνωσης σεμιναριών για δημοσιογράφους από όλες τις χώρες μέλη και αυτό για πολλά νομοθετικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί για τον κανονισμό και την οδηγία όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους δημοσιογράφους είτε επειδή έχουν προσωπικό ενδιαφέρον, είτε για τη δουλειά τους, να μπορούν να έρχονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενημερώνονται για τη δουλειά που γίνεται εδώ και να τους δίνεται η ευκαιρία να συζητούν με τους Ευρωβουλευτές που είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα νομοθετικά μέτρα. Θέλω να σας πω επίσης ότι η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μοναδική γιατί δουλεύουμε με 22-23 πιο σωστά γλώσσες από τον Ιούλιο τουλάχιστον, αφού έχουμε και την Κροατία μεταξύ μας. Είναι, πιστεύουμε, πολύ σημαντικό και για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και για τους πολίτες στα κράτη-μέλη να μπορούν το μήνυμά μας να το παίρνουν στη γλώσσα τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, όπως γνωρίζετε, είναι ένας πολυπολιτισμικός οργανισμός και πολυγλωσσικός με, που αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια πολιτών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Τέλος, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι του χρόνου, το 2014, στις 22 και 25 Μαΐου του χρόνου, θα έχουμε τις επόμενες ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές πολύ σημαντικές αυτή τη φορά. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντικές γιατί τώρα που έχει αρχίσει ήδη να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες στα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει από κοινού με τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου για το 95% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι εκλογές αυτές έχουν και μια άλλη διαφορά. Το αποτέλεσμα θα παίξει σημαντικό ρόλο για την εκλογή του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον διάδοχο δηλαδή του κ. Μπαρόσο. Οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων δηλαδή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των επόμενων ευρωεκλογών για να προτείνουν τον επόμενο πρόεδρο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες στην Ευρώπη σήμερα συζητούν, διαπραγματεύονται και θα αποφασίσουν τελικά ποιος θα είναι ο υποψήφιος που θα προτείνουν. Οι εκλογές αυτές λοιπόν είναι διαφορετικές, σημαντικές, γιατί δεν θα είναι εκλογή για διαφορετικές ιδέες και προγράμματα, αλλά και για διαφορετικές προσωπικότητες. Αυτά προς το παρόν. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Ελπίζω να έχετε ενδιαφέρουσα διαμονή εδώ στις Βρυξέλλες και να βρείτε και το σεμινάριο αυτό πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα σας δείξουμε ένα μικρό φιλμάκι για την υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο θα δείτε τι προσφέρουν, τι προσφέρει η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους δημοσιογράφους όπως είσαστε εσείς.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 θα σας παρουσιάσει κάπως σύντομα το πρόγραμμα του σεμιναρίου μας αυτού και θα σας δώσει και κάποιες πληροφορίες για την εκστρατεία μας όσον αφορά την προστασία δεδομένων, τον κανονισμό και την οδηγία. Όλα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια απεργία στο Ζάβεντεμ και ίσως αυτό να δυσκολεύει ορισμένους να φτάσουν. Ελπίζω να μην αργήσουν πολύ. Να σας δώσω κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα ότι έχετε διερμηνία. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και ισπανικά. Μπορείτε λοιπόν και να μιλάτε σε αυτές τις ε, γλώσσες, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, αλλά και να τις ακούτε. για το σεμινάριο τώρα. Πρώτα θα έχουμε μια γρήγορη εισαγωγή όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσουμε πώς βοηθούμε τους ευρωβουλευτές να ετοιμάζουν τις εκθέσεις τους, τις προτάσεις τους. Αυτό είναι κάπως άτυπο το κομμάτι. Μετά Όλα τα υπόλοιπα είναι on record. Το πρώτο κομμάτι είναι off the record. Θα υπάρξουν και Twitter. Θα δείτε ότι θα υπάρξουν διάφορες ερωτήσεις, απαντήσεις. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να παρέμβετε. Σήμερα το απόγευμα ουσιαστικά έχουμε συζήτηση μεταξύ μας για την προστασία δεδομένων με τους διάφορους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα από διάφορες οργανώσεις. Ενώ αύριο θα έχουμε εδώ και τον επόπτη προσωπικών δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τους ευρωβουλευτές, εκείνους που στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές εκπονούν τις σχετικές προτάσεις και εκθέσεις. Θα σας πω δύο λόγια λοιπόν πρώτα απ' όλα τι γίνεται με την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ρόλο παίζουμε εμείς. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις πρώτα απ' όλα προς τους δημοσιογράφους. Είναι διάφορες αυτές, μία από αυτές είναι η προστασία δεδομένων. Και στην περίπτωση αυτή προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσουμε απευθείας και με τον Ευρωπαίο πολίτη. Υπάρχουν κάποια μέσα για τις ανακοινώσεις μας που χρησιμοποιούμε, ο συνάδελφος Deutsche θα σας πει περισσότερα και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να τα γνωρίζετε για να μπορείτε και να τα χρησιμοποιήσετε εφόσον κάποια στιγμή σας φανεί αυτό χρήσιμο. Ο Γιάννης έλεγε να, ότι ο συνάδελφος εκεί είναι εντυμένη στα κίτρινα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Επίτηδες έχει εντυθεί στα κίτρινα γιατί ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η αστερίσκη που θα έχετε δει και στα έγγραφα που πήρατε. Το είχε πει λοιπόν ότι θα ντεθεί στο ίδιο χρώμα με τα αστέρια αυτά για να ενισχύσει ακριβώς την δράση μας. Τι θέλουμε να δείξουμε με αυτό. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα αλλά πίσω από αυτά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, υπάρχει δουλειά που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μικρά γράμματα πολλές φορές που δεν διαβάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να συνειδητοποιήσετε ότι το τελικό αποτέλεσμα της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων Φερρυπίν αποτελεί τον καρπό μιας μακράς κοινοβουλευτικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε ακούσει όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις, εξού και ο αστερίσκος, ο κίτρινος αστερίσκος που βλέπετε. Ο συνάδελφος Ντότσε θα σας αναφέρει τα άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μια πολύ σημαντική στιγμή στη διαδικασία θα είναι η ψηφοφορία στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο ή κάπου εκεί. Μιλάμε για την προστασία δεδομένων σήμερα. Θα σας δείξουμε αν ε, είμαστε έτοιμοι τεχνικά την συνολική ιδέα. Έχουμε έρθει σε επαφή με τρεις επαγγελματίες, επαγγελματίες ενώ για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη και απόλυτη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν οι νομικοί, οι οποίοι εξετάζουν το θέμα και φυσικά βάζουν ε, τα δικά τους ε, στοιχεία αλλά αυτοί οι όροι που βάζουν οι νομικοί στις διάφορες συμφωνίες συνήθω γράφονται με τα ψηλά γράμματα, είναι τόσο πολύπλοκοι και θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι δεν τα διαβάζουμε καν. Ε, το δεύτερο επαγγελματικό κλάδο είναι εκείνο που ασχολείται με το λεγόμενο profiling, δηλαδή με την ε, συγκέντρωση ε, γνωρισμάτων σχετικά με αυτόν που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Έτσι, συλλέγουν οι επαγγελματίε αυτή τα δεδομένα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προσώπου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ανάλογα το στέλνουν διαφημίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και έπειτα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον ιδιωτικό σα ε, βίο με εγκληματικό τρόπο, οι hackers. Δεν αποτελεί φυσικά μέρος της νομοθεσίας αυτής καθεαυτής, αλλά η συλλογή πολλών προσωπικών δεδομένων σίγουρα οδηγεί μερικές φορές σε καταχρήσεις. Έχουμε λοιπόν έρθει σε επαφή με αυτά τα τρία ίδια επαγγελματιών. Τους ζητήσαμε να μας δώσουν ε, κάποια, κάποιες συμβουλές και να. Α, είναι έτοιμο το βίντεο. Βάσει αυτών των τριών βίντεο καταλήξαμε και σε αυτό που έχετε και στα χέρια σας, που είναι ένα μικρό εγχειρίδιο, στο οποίο αναφέρονται 10 συμβουλές για να προστατεύσετε το προσωπικό σας βίο στο διαδίκτυο. Μετά θα μιλήσουμε βέβαια για το θέμα από την πλευρά και την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπες για την προσέγγιση αυτών των ε, μικρών ταινιών. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Στο χέρι μας είναι να προστατευτούμε. Αλλά δεν φτάνει, συμφωνώ. Και γι' αυτό χρειάζεται και νομοθεσία. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του εγχειριδίου αυτού που έχετε στα χέρια σας. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε παραπάνω και ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείται η νομοθεσία. Και εκεί είναι που παρεμβαίνουν οι ευρωβουλευτές και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας πρέπει να εξυγχρονιστεί και να λάβει υπόψη της τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στον τομέα του διαδικτύου για να μπορεί να βοηθήσει αυτή η νομοθεσία.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 So, Καλώς, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι που μας παρουσιάσατε την εκστρατεία μας. Τώρα, πριν περάσουμε στο πρώτο τμήμα του προγράμματος, επιτρέψτε μου να σας πω και κάποιες πληροφορίες για την νομοθετική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, πώς λειτουργεί αυτή. Και αυτό για να καταλάβετε κάπως καλύτερα τι ακριβώς συζητάμε και πώς η νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε πρόκειται για κανονισμό, είτε πρόκειται για οδηγία, υιοθετείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μια και από το Συμβούλιο των Υπουργών από την άλλη. Μερικοί από εσά είσαστε ήδη εξοικειωμένοι με αυτές τις διαδικασίες, άλλοι όχι. Γι' αυτό λοιπόν, συγγνώμη ζητάω από τον προτέρων από τους συναδέρφους που τα ξέρουν όλα αυτά, ξέρουν ποιε είναι οι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά για τους άλλους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν αρκετά καλά θα είναι χρήσιμο φαντάζομαι. Συνεπώς, αρχίζουμε με αυτή την PowerPoint παρουσίαση. Όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ μιλάμε για έναν κανονισμό και για μία οδηγία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας εξηγήσω αυτά τα δύο είδη νομοθετημάτων πώς εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ρόλο παίζουν δηλαδή για την έγκριση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στην υιοθέτηση ακριβώς των νομοθετημάτων αυτό. Λοιπόν, να, εδώ βλέπετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάνω, η οποία έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας να προτείνει μια νέα νομοθεσία. Η Επιτροπή δηλαδή στέλνει και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ένα πρώτο σχέδιο μιας πρότασης για νομοθεσία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει και το προσχέδιο προπολογισμού. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει στους 754 απευθείας με καθολική ψηφοφορία εκλεγμένους ευρωβουλευτές και συγχρόνως πηγαίνει και στο Σεβούλιο Υπουργών, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς των 27 χωρών μελών. Ε, ποιοι υπουργοί? Οι υπουργοί, οι αρμόδιοι που έχουν το χαρτοφυλάκιο δηλαδή, το σχετικό με το θέμα το οποίο προτείνεται ως νομοθεσία. Επιτρέψτε. Να σας δώσω τώρα και λίγες πληροφορίες πώς χωρίζονται στο Κοινοβούλιο οι έδρες αναχώρα. Όπως βλέπετε, ίσως η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο αριθμό εδρών που ανέρχεται σε 99 για την ώρα. Χώρες όπως Εσθονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος έχουν έξι βουλευτές, έξι έδρες. Όλα αυτά βέβαια θα αλλάξουν μετά από την ένταξη της Κροατίας που προβλέπεται τον Ιούλιο και θα αναθεωρηθούν άλλη μια φορά στις επόμενες ευρωεκλογές. όπου θα εκλεγούν 751 ευρωβουλευτές. Οι κύριοι φορεί τη δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτικέ ομάδε. Είναι δηλαδή μεγάλε πολιτικέ οικογένειε που εκπροσωπούν τι μεγάλε πολιτικέ τάσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη πολιτική ομάδα, ε, σε δύναμη δηλαδή, είναι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, που εκπροσωπεί τη συντηρητική και χριστιανοδημοκρατική πλευρά του πολιτικού φάσματος στην Ευρώπη. Ακολουθούν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, δηλαδή της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, που είναι η δεύτερη σε δύναμη και ε, ανέρχονται σε 100, 190 οι πρώτοι είχαν 270, μετά είναι φιλελεύθεροι, πράσινοι Υπάρχει και η ομάδα που λέγεται ECR, δηλαδή μια ομάδα που εκπροσωπεί ευρωσκεπτιστικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαρτίζεται κυρίως από Βρετανούς συντηρητικούς. Ακολουθεί η αριστερά, η Γκουε, δηλαδή η ενωτική αριστερά, στην οποία εκπροσωπούνται οι γερμανικοί Λίνκε αλλά και κομμουνιστικά κόμματα και ούτω καθεξής. Και τέλος το EFD Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας που και αυτό έχει ε, αρκετά ευρωσκεπτικιστική ε, τοποθέτηση. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 20 διαρκείς επιτροπές όπως και κάθε κοινοβούλιο στον κόσμο άλλωστε χωρίζεται δηλαδή σε επιτροπές ε, το έργο του έχει κοινοβουλευτικές επιτροπές επομένως αρμόδιες για διάφορους τομείς της νομοθεσίας με διαφορετικές αρμοδιότητες, για παράδειγμα η Επιτροπή Μεταφορών, αρμόδια για θέματα μεταφορών, ασφάλειας μεταφορών και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την προπαρασκευή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αυτή των των ε, ε, θεμελιωδών ελευθεριών εσωτερικών και δικαιοσύνης. Αύριο θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις με μέλη της Επιτροπής αυτής, δηλαδή με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Τι θα πούν αυτά τα λόγια τώρα. Είναι βέβαια κάπως η ειδική τεχνική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν η Κομισιόν καταθέτει πρόταση νόμου αυτό διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αρμόδια δηλαδή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία καθορίζει έναν εισηγητή, που είναι ο κύριος υπεύθυνο για την σύνταξη της θέσης του Ευρωκοινοβουλίου. Στο έργο του τον βοηθούν οι λεγόμενοι σκιώδεις εισηγητές, που είναι αυτοί που εκπροσωπούν τις άλλες πολιτικές ομάδες. Επίσης, πολύ σύντομα, κάποια στοιχεία για την νομοθετική διαδικασία ή τις νομοθετικές διαδικασίες. Έχουμε την συνδιαλλαγή, τη διαβούλευση, συγγνώμη, τη διαβούλευση που έχει περιοριστεί πια σε πολύ περιορισμένο τμήμα της νομοθεσίας μετά από την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη που εφαρμόζεται ιδίως σε διεθνείς συμφωνίες τις οποίες υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες του κόσμου, όπου το Κοινοβούλιο έχει την, την δυνατότητα μόνο να εγκρίνει ή να απορρίψει τη συμφωνία. Και τέλος, αλλά και πιο σημαντική, η διαδικασία συναπόφασης ή τακτική νομοθετική διαδικασία, η συνήθις νομοθετική διαδικασία, όπως αποκαλέστηκε μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, που είναι κατά κάποιο τρόπο αυτή που καλύπτει ε, στην ουσία το μεγαλύτερο φάσμα τη ε, νομοθετική δραστηριότητα. Εκεί το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει την προτινόμενη νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να την απορρίψει ή να την τροποποιήσει. Κάτι το οποίο βεβαίω συμβαίνει και συνήθω. Τέλο, λίγα λόγια, λίγε πληροφορίε σχετικά με την συναπόφαση και τα διαφορετικά βήματα τη διαδικασία αυτή. Όπω σα είπα και στην αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θεσμικό εκείνο όργανο το οποίο διαθέτει το δικαίωμα πρωτοβουλίας να καταθέτει δηλαδή νομοθετικές προτάσεις, σχέδια νόμων τα οποία υποβάλλει ή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο Συμβούλιο των Υπουργών και αυτοί οι δύο θεσμοί μετά καλούνται να συμφωνήσουν επί της νομοθεσίας. Αυτό μπορούν να το πράξουν και σε μια πρώτη ανάγνωση αν δεν συμφωνήσουν θα προχωρήσουν σε δεύτερη ανάγνωση και εάν ακόμη δεν συμφωνήσουν τότε προχωρούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής, conciliation procedure. Εάν συμφωνήσουν ή όταν συμφωνήσουν, καταλήγουν στο, στην νομοθετική πράξη, την οποία υπογράφει και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή το Συμβούλιο, και εάν δεν συμφωνήσουν βέβαια χρειάζεται πλέον να ανακληθεί, η, να αποσυρθεί η ε, νομοθετική πρόταση και να υποβληθεί νέα. Έτσι έχει κάπως η διαδικασία, αν και βέβαια είναι αρκετά λαβύρινθος ακόμα και για τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι λίγο δύσκολο να την αντιληφθεί, να την αφομοιώσει κανείς. Αν έχετε όμως ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις θέσετε αμέσως τώρα. Αν δεν έχετε, να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Καλό σας απόγευμα και ελπίζω και εύχομαι οι συζητήσεις σας να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. you see the screen? Την ε, οθόνη τη βλέπετε? Δεν την καλύπτουμε εμείς που καθόμαστε εδώ μπροστά, όχι. Ναι, τη βλέπετε ωραία. Τώρα, να προχωρήσουμε στον φάκελο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λυσμονήσαμε να σας πούμε πριν ότι αν και αυτό βέβαια είναι θέμα ε, διαδικτύου, έχουμε παραγγείλει και μερικά ε, μπλοκ, οπότε ίσως αν θέλετε να τα χρησιμοποιήστε, να γράψετε. Γιατί μπορείτε να γράψετε πολλά από αυτά που θα πούμε το διήμερο. Είμαι βεβαία ότι θα σας δώσουμε πολλές ε, ε, πληροφορίες. Είμαι βεβαία ότι θα σας φανούν χρήσιμα τα ε, μπλοκ αυτά. Προχωρούμε τώρα να σας παρουσιάζω το πάνελ. Αυτό το μέρος εδώ είναι off the record, όπως είπα και πριν. Εδώ δεξιά μου είναι η Νατάλια Ντασίλβα, Έχουμε αρκετούς Ισπανούς εδώ πάνω τώρα. Νατάλια Ντασίλβα, Ισπανίδα και αυτή και press officer του Κοινοβουλίου, επίσημη press officer δηλαδή, και παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Αριστερά μου είναι ο Χωσέ Μανουέλ Ντεφρούτος, πάλι Ισπανός, και είναι ο αξιωματούχος της Επιτροπής που επεξεργάζεται την νομοθεσία αυτή. Να δώσω πρώτα το λόγο στην Αταλία να σας κάνει μια σύντομη εισαγωγή στον φάκελο και μετά να συμπληρώσει ο Χωσέ Μανουέλ και να μας μείνει χρόνος ελπίζω για ερωτήσεις γιατί θα έχουμε περίπου 45 λεπτά συνολικά. Ευχαριστώ όπως σας εξήγησε, θα σας πω λίγα λόγια για την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση της ε, προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων και μετά ο Χωσέ Μανουέλ θα σας, πω, πει περισσότερα πράγματα, περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, να σας δώσω λίγο τη γενικότερη ιδέα της μεταρρύθμισης σε αυτήν εδώ την πρώτη διαφάνεια που βλέπετε. Έχουμε ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα έχουμε μια οδηγία του 1995 καθώς και απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου του 2008. Η οδηγία είναι πιο γενική και η απόφαση πλαίσιο είναι πιο συγκεκριμένη, πιο ειδική. Αναφέρεται κυρίως σε αστυνομική και δικαστική συνεργασία για ποινικά θέματα. Τώρα, στην τρέχουσα οδηγία προβλέπεται νέα νομοθεσία, νέα γενική νομοθεσία με στόχο να προσαρμοστούν οι αρχές που περιλαμβάνονται στην ήδη ισχύουσα ε, νομοθεσία, οδηγία δηλαδή, να προσαρμοστούν λοιπόν οι αρχές αυτές στο διαδίκτυο και σε άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, διότι βέβαια η οδηγία του 1995 δεν είναι πλέον επίκαιρη από την άποψη αυτή. Και αυτό θα καλύψει πιο, τα, πιο πολλές πτυχές του data processing και online και offline. Δηλαδή μηχανές αναζήτησης, αρχεία νοσοκομείων, αρχεία ε, πανεπιστημίων και οτιδήποτε τέλος πάντων επεξεργασία δεδομένων. Στη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης που άρχισε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως υποχρεούται όταν ε, πρόκειται να υποβάλει την πρόταση αναθεώρησης ήρθε σε επαφή με διαφόρους ενδιαφερομένους με τον κλάδο, με ακτιβιστές και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από την υποβολή της μεταρρύθμισης αυτής, τον Ιούλιο του 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε θέση σχετικά με το περιεχόμενο της μελλοντική αυτής μετα, μεταρρύθμισης. Στην έκθεση ΒΟΣ, όπως βλέπετε γραμμένο εκεί. Ψήφισμα λοιπόν, στο οποίο κατέληξε η έκθεση αυτή, με κύριο μήνυμα ότι οι αρχές που θεσπίζει η τρέχουσα οδηγία το 1995 αποτελούν το σημείο αφετηρίας και πάνω σε αυτές τις αρχές πρέπει να βασιστεί και παραπέρα προσαρμογή ή μεταρρύθμιση. Σε αυτή την πρώτη διαφάνεια στοχεύουμε να σας δώσουμε μια επισκόπηση για τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης έτσι ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο οι ίδιοι οι άνθρωποι. Προσαρμόζονται δηλαδή, προσαρμόζονται οι κανόνες στη νέα εποχή του διαδικτύου. Παρακολουθούνται έτσι οι τεχνολογικές εξελίξεις, διότι καμιά φορά ο κόσμος έχανε τον έλεγχο των δεδομένων του, ιδίω επιγραμμικά, online. Έτσι λοιπόν, η ιδέα είναι ο άνθρωπος, το άτομο, να έχει έλεγχο, να γνωρίζει ακριβώς τι δεδομένα δίνει και σε ποιον. Δεύτερο στόχος ήταν να υπάρξει πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού, διότι καμιά φορά μια ευρωπαϊκή εταιρεία που θέλει να αρχίσει να λειτουργεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς κανόνες, κανονισμούς, νομοθεσία της άλλης χώρας. Έτσι λοιπόν η οδηγία θα βάλει ένα ελάχιστο επίπεδο προδιαγραφών. Αλλά μετά κάθε χώρα μέλος μπορεί να αποφασίσει αν θα βάλει παραπέρα στάνταρτ, παραπέρα προδιαγραφές ή πιο αυστηρές ενδεχομένως. γιατί ήταν μια έξτρα δυσχέρεια για τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, γιατί και κόστος συνεπήγε το αυτό και βεβαίως χρειαζόταν και χρόνο και ιδιαίτερη προσπάθεια εφόσον ήθελαν να κινηθούν διεθνώς. Τέλος, οι βασικοί ευρωβουλευτές με τους οποίους θα μιλήσετε αύριο είναι ο Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ, Γερμανός από τους Πράσινους. Αυτός είναι ο βασικός εισηγητής, αρμόδιος δηλαδή για τη σύνταξη του κειμένου του Γενικού Κανονισμού. Και ο Δημήτριος Δρούτσας, σοσιαλιστής, Έλληνας και σκιώδης εισηγητής για την ομάδα του. Προχωρώ στη δεύτερη διαφάνεια, όπου βλέπετε μερικές βασικές ημερομηνίε. Τι έγινε και τι θα γίνει στο Κοινοβούλιο μετά από την κατάθεση πρόταση της Κομισιόν. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2013. Αντέδρασαν οι εισηγητές που σας ανέφερα προηγουμένως, Άλβρεχτ και Δρούτσας, με κατάθεση τροπολογιών πάνω στο κείμενο της Κομισιόν. Μετά πήγε στις διάφορες ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου, δηλαδή κυρίως απασχόλησης, βιομηχανίας. Ένα λεπτό να βρω νομικές υποθέσεις και ενιαίας αγοράς, εσωτερικής αγοράς δηλαδή και προστασίας καταναλωτή οι οποίες ε, επιτροπές καταθέτουν γνωμοδοτήσεις παρόλο που δεν είναι οι καταρχήν ας πούμε αρμόδιες επιτροπές που είναι η Επιτροπή των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Αυτά μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Τώρα, Μάρτιο-Ιούνιο γίνονται οι συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και ο στόχος είναι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ε, ομάδων που να καλύπτει και την οδηγία και τον κανονισμό πριν από τι θερινέ διακοπέ. ώστε να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών πριν από τον Ιούλιο, 7ο δηλαδή. Και η ψηφοφορία αυτή θα δώσει στου δύο εισηγητέ που διορθώνει ο Ιδρυνέας, είναι και οι δύο ισο, ισότιμοι, ισοδύναμοι, δεν είναι σκιώδη ο κ. Δότσα, έχει τον κανονισμό, ώστε μετά να μπορέσει να προχωρήσει και στο Συμβούλιο για να καταλήξουν όλες οι χώρε μέλη σε συμφωνία. Αυτό θα γίνει το δεύτερο μισό του 2013. Αν όλα πάνε καλά, η τελική ψηφοφορία για το κείμενο θα γίνει αρχές του 2014. Πρώτα στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών και μετά θα ακολουθήσει στην Ολομέλεια. Στην τρίτη τώρα διαφάνεια αν θέλετε να προχωρήσετε παρακαλώ στο τρίτο slide, στην τρίτη διαφάνεια, μερικά νούμερα που μπορεί να σας φαίνονται ενδιαφέροντα. Δηλαδή τι εύρος έχει αυτή η νομοθεσία. Καθημερινά χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην Ευρώπη 250 εκατομμύρια άνθρωποι. Ακούσατε για τις τροπολογίες που είναι σχεδόν 4.000 τροπολογίες για τον γενικό κανονισμό. 3.999 τροπολογίες. Συνολικά, στα πλαίσια της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, αλλά εφόσον λάβει κανείς υπόψη και τις συνεισφορές των υπόλοιπων επιτροπών. 771 τροπολογίες έχουν κατατεθεί για την οδηγία. Όταν κατέθεσε την πρότασή της η Κομισιόν είπε επίσης ότι ότι θα εξοικονομούσαν οι διάφορες επιχειρήσεις συνολικά μέχρι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο εφόσον θα μπορούσαν να βασιστούν σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Να μην χρειάζεται δηλαδή να ε, προσαρμόζονται σε διαφορετικούς κανόνες εφόσον κινούνται διεθνώς. Επίσης εξοικονόμησε 130 εκατομμυρίων ευρώ από την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας χάρη στην αναθεώρηση αυτή. Και σύμφωνα και με ένα ευρωβαρόμετρο, το οποίο πάλι υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όταν ε, κατέθεσε δηλαδή την μεταρρύθμιση, 70% των Ευρωπαίων ανησυχούν για ενδεχόμενη κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων τους. 72% των ε, χρηστών διαδικτύου στην Ευρώπη ανησυχούν διότι θεωρούν ότι τους ζητούν υπερβολικά πολλά δεδομένα στο ε, διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ο Μανουέλ τώρα. Μας μιλήσει και αυτός για κάποια σημεία της πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. Θα, θα προσπαθήσω κάπως σύντομα να σας παρουσιάσω το στόχο και το νόημα της τροποποίησης αυτής της αναθεώρησης των ρυθμίσεων που υπάρχουν για την προστασία δεδομένων. Και θα σας πω και ποια είναι η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα κάνω αυτό σύντομα για να μπορέσουμε και να συζητήσουμε μετά. Το πρώτο λοιπόν που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι ποιο είναι το σημερινό πλαίσιο που έχουμε για την προστασία δεδομένων, το νομικό πλαίσιο. Έτσι. Έχουμε ήδη διάφορα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πιο σημαντικό είναι η οδηγία του 95 αριθμός 46 που υιοθετήθηκε το 95 και που θέτει το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων στις διάφορες χώρες και καλύπτει και τις online δραστηριότητες και τις άλλες. είτε πρόκειται για ασφαλιστικές εταιρείε, είτε πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε για οτιδήποτε. Μετά έχουμε την οδηγία 58 του 2006 που αναφέρεται πιο πολύ στις τηλεπικοινωνίες. Μετά έχουμε τον κανονισμό πρέπει να ξέρουμε ότι η οδηγία έτσι καλώς εφαρμόζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και καλύπτει δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία δεδομένων από οποιονδήποτε πλην των αρχών που εφαρμόζουν τον νόμο, που επιβάλλουν τον νόμο. ο, η απόφαση πλαίσιο του 2008-977 προσπάθησε να κάνει κάποια εναρμόνιση για την επεξεργασία δεδομένων, χωρίς να πρόκειται βέβαια για πλήρη εναρμόνιση. Απλώς θέτει κανόνες και για τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικές δραστηριότητες. Έπειτα έχουμε άλλα μέσα που είναι το Schengen, η Europol, η Eurojust, Eurodac κλπ. και, Και αυτό σας τα λέω για να καταλάβετε ότι η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα επιμέρους ζητήματα δεν συντονίζονται πάντα αρκετά καλά Η παρουσία αποτελείται από τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, γιατί αλλάζουμε τους κανόνες για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ποιοι είναι οι στόχοι της πολιτικής που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ε, τρίτον, τι περιλαμβάνει το πακέτο για την μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων. Και μετά θα σας μιλήσω για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα για την μεταρρύθμιση. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τους υπάρχοντες κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παρουσιάσει ένα νέο πακέτο προτάσεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Γιατί? Γιατί θέλει να καλύψει διάφορες αλλαγές, διάφορες εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά τις αλλαγές που είχαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2005 και μετά είτε πρόκειται για τη χρήση του διαδικτύου, είτε πρόκειται για συμφωνίες διεθνείς, είτε πρόκειται για διαφορετικό τρόπο λήψη αφάς κλπ. κλπ. Έπειτα υπάρχουν θεσμικές αλλαγές. Μέχρι τώρα είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει το άρθρο 16 που λέει ότι η προστασία δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η επεξεργασία δεδομένων γίνεται με εποπτεία από αρμόδιες αρχές και υπό όρους μόνο. Έπειτα έχουμε και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο άρθρο μιλάει για την προστασία προσωπικών δεδομένων και λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον προσωπικό βίο. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί τώρα έχουμε νέα νομική βάση και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καλύψει με το νέο αυτονομικό σύστημα όλες τις περιπτώσεις προστασία προσωπικών δεδομένων. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δει τι ειδικά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα ή επιχειρήσεις μετά από το 1995 και τη θέση ισχύ της προηγούμενης οδηγίας, δηλαδή τι κενά παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή γιατί μην ξεχνάμε ότι οδηγία σημαίνει ότι πρέπει να ενσωματωθεί από 27 διαφορετικά νομοθετικά συστήματα, σε 27 δηλαδή διαφορετικέ χώρε. Άρα ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η ενσωμάτωση αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και έτσι μερικέ φορέ οι διατάξει τη σχετική νομοθεσία σε μία χώρα μπορεί να προστατεύει περισσότερο από ό,τι σε μια άλλη. Και υπάρχουν διαφορές. Λοιπόν, άρα και για τις επιχειρήσεις και για τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την επεξεργασία των δεδομένων, η ζωή τους γίνεται πάρα πολύ δύσκολη αφού ισχύουν διαφορετικοί νόμοι, διαφορετικές ρυθμίσεις σε διαφορετικές χώρες. Άλλος λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να δει λιγάκι πώς εφαρμόζεται η προστασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου. Ξέρουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούνται σήμερα από τις αρχές επιβολής του νόμου για να βοηθούν στην πρόληψη τρομοκρατικών ε, επιθέσεων. Χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, άρα στοιχεία οικονομικά επίσης. Προκειμένου λοιπόν όλες αυτές οι πτυχές να αντιμετωπιστούν, αποφάσισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία νέα πρόταση το 2012. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι της πολιτικής με τη μεταρρύθμιση αυτή. Είναι απλή. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θέλουν να ενισχυθούν οι δυνατότητες προστασίας. Θέλουν επίσης να υπάρξει ένα νέο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Επίσης η πρόταση θέλει να έχει πιο ισχυρές θεσμικές ρυθμίσεις και να συνεισφέρει στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως δεν θέλει να φτιάξει ένα νέο σύστημα προστασίας δεδομένων, διαφορετικό εντελώς από το τρέχον σύστημα. Η πρόταση που ήδη ξεκίνησε από το 2011 είναι στο πλαίσιο και στην οδηγία δηλαδή το 95 να προσθέσει στοιχεία για να βελτιωθεί το νομικό σύστημα και να καταργηθούν τα προβλήματα ή τα ζητήματα τα οποία είχαμε αντιμετωπίσει στα 15 χρόνια που ίσχυε η προηγούμενη οδηγία να αντιμετωπιστούν όλες οι δυσκολίες που έχουν αναφερθεί δηλαδή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία μέχρι σήμερα. Τώρα το πακέτο αποτελείται από δύο νομικά μέσα. Υπάρχει ο κανονισμός, ο οποίος καθορίζει την ομοθεσία για την γενική προστασία δεδομένων στα κράτη-μέλη, από τα κράτη-μέλη και από οποιονδήποτε ασχολείται με επεξεργασία δεδομένων εκτός από τις αρχές επιβολής του νόμου. Αν πρόκειται για επιβολή νόμου, τότε το θέμα αυτό καλύπτεται από άλλη ρύθμιση. Πρόκειται λοιπόν για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε άλλο εκτός από την επιβολή του νόμου στις ε, χώρες μέλη, επεξεργασία δεδομένων κλπ. για να αντιμετωπιστούν, όπως είπαμε, τα κενά από προηγούμενες ρυθμίσεις. Με τον κανονισμό, σύντομα όπως σας είπα, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο για συζήτηση, ο κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία του 1995, συνεχίζει να προστατεύει την, τα δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός, δεν είναι πιο οδηγία, είναι κανονισμός, θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες, χωρίς να χρειάζεται η κάθε χώρα ξεχωριστά να ενσωματώσει την νομοθεσία στο... με διαφορετικό τρόπο δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει καλύτερη ομοιομορφία και οι χώρες και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε κάθε χώρα θα γνωρίσουν έτσι πολύ καλύτερα ε, πώς πρέπει να εφαρμόσουν τη ρύθμιση αυτή. Ενισχύεται η προστασία δεδομένων των ατόμων. Αυτό είναι πολύ βασικό. Υπάρχει πιο ξεκάθαρη ενημέρωση προς τους Ευρωπαίους πολίτες διευκολύνεται η περιγραφή των διαφόρων δικαιωμάτων, το δικαίωμα ε, στο να μπορεί να ξεχαστεί κάποιος, πότε μπλοκάρουν τα προσωπικά δεδομένα κλπ. κλπ. Υπάρχει ένα σύστημα κοινοποίησης Και το άλλο σημείο που θίγεται εδώ πέρα είναι η συνένεση που δίνει ο χρήστη του διαδικτύου για να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, η οποία πρέπει να είναι ρητή και να μην υπονοείται απλώ. Στόχος μας είναι δηλαδή όλα αυτά να ευθυγραμμιστούν καλύτερα προς την ιδέα της ενιαίας αγοράς. Διάλο βασικά στοιχεία του κανονισμού είναι η διαχείριση των δεδομένων, αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό ήδη. Ο κανονισμός θα βοηθήσει τις αρμοδιότητες, αρμοδιότητες των εποπτών προσωπικών δεδομένων, που είναι ανεξάρτητες αρχές, θα υπάρχει πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υφόρων εποπτών για την εφαρμογή του κανονισμού, καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρχών και συνεργασία και θα υπάρχουν και μηχανισμοί που θα διευκολύνουν τη συνεργασία αυτή συγκεκριμένη. Θα υπάρχουν και ρυθμίσεις για τη διεθνή διάσταση του ζητήματος. Δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διεθνές. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει και με εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και από τις τρίτες χώρες και επίσης να έχουν το δικαίωμα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύονται ακόμα και όταν πρόκειται για παραβιάσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Το δεύτερο μέσο για την ε, προστασία δεδομένων για την ε, αστυνομία και ως εξής. Είναι μια οδηγία η οποία αντικαθιστά την ε, συμφωνία πλαίσιο. Προσπαθεί να καλύψει και το εθνικό επίπεδο. Σήμερα πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο όταν πρόκειται για δεδομένα στα οποία μπλέκονται δύο χώρες. Όταν πρόκειται για μία μόνο χώρα δεν υπάρχει μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς το παρόν για να υπάρχει αυτή η προστασία προσωπικών δεδομένων. Ενώ με την οδηγία αυτή υπάρχει και αυτή η κάλυψη. Η οδηγία αυτή θα επεκτείνει τις αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό και σε αυτή την περίπτωση με βέβαια κάποιους περιορισμούς που επιβάλλονται λόγω των δραστηριοτήτων της αστυνομίας ή άλλων αρχών επιβολής του νόμου. Και περνάω στο τελευταίο μέρος τώρα. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η συναπόφαση. Η Επιτροπή Ελευθεριών του νομου και περνω στο είναι η επί της ουσίας αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που ετοιμάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συγητές είναι ο κύριος Άλμπρεχτ και ο κύριος Δρούτζας. Οι άλλες επιτροπές γνωμοδοτούν. Είδαμε πώς λειτουργούν όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ε, τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο ετοιμάστηκαν τα πρώτα έγγραφα, έγιναν ε, τα σχέδια εκθέσεων από τους εισηγητές Τώρα είμαστε στη διαδικασία που συζητιώνται οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί τόσο στον κανονισμό όσο και στην οδηγία. Ε, είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες όπως είπαμε και στον κανονισμό και στην οδηγία. Οι εισηγητές με τις πολιτικές ομάδες εργάζονται σκληρά προκειμένου να ετοιμάσουν κάποιους συμβιβασμούς για να μπορέσει τελικά να εγκριθεί και το κείμενο. Στο Συμβούλιο τώρα. Και εκεί δουλεύουν σκληρά υπό την Ιρλανδική Προεδρία, προκειμένου και εκεί να καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό. Και η δικιά του συμφωνία θα έρθει στο Κοινοβούλιο, η δικιά μας ε, στο Συμβούλιο και τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε μεταξύ μας, οι συνομοθέτες δηλαδή, για να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία πάνω στο πακέτο αυτό. Πριν το τέλος της θητείας αυτής ελπίζουμε. Θα παραμείνω εδώ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, ευχαρίστως να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα μας μένει λίγος χρόνος για ερωτήσεις. Αν έχετε λοιπόν ερωτήσεις, όπως είπα πάντα εδώ είναι off the record, πέστε το όνομα καθώς και το μέσο για το οποίο εργάζεστε. Μπορούμε να ακούσουμε όλων των ειδών τι ερωτήσει. Αν θέλετε τώρα ερωτήσεις, να κάνετε ερωτήσει για να πάρετε απόψει, αυτό καλύτερα το αφήστε για του ευρωβουλευτέ στο δεύτερο μέρο τη ε, συνάντηση. Είμαι freelance και εργάζομαι σε διάφορα σκανδιναβικά media. Με ενοχλεί η προτινόμενη οδηγία γιατί να καλυφθούν και οι εγχώριες μέσα στις χώρες, δηλαδή ροές ε, των ε, δεδομένων. Μπορείτε να δώσετε κάποια απάντηση σε αυτό. Χωσέ Μανουέλ, όπως σας είπα, σήμερα στην αρχιτεκτονική της προστασίας των δεδομένων υπάρχουν ειδικοί κανόνες δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για ε, θέματα law enforcement, δηλαδή αστυνομίας, δικαστικά κτλ. Έχετε τώρα κανόνες για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο διαφορετικών αστυνομιών, ας πούμε. Όμως, η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Επομένως, βεβαίως, μεταξύ χωρών μελών. Τώρα, για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα γίνεται σεβαστό σε όλες τις περιστάσεις, δηλαδή και εγχωρίως, χρειάζεται κάποιος συντονισμός. Εφόσον η αστυνομία διαθέτει κάποιο δεδομένο ενός προσώπου σχετικά με κάποια ποινική δίκη ή έρευνα ή ανάκριση. Δεν μπορείτε να ξέρετε από την αρχή εάν η χρήση του δεδομένου θα είναι μονάχα εθνική ή θα ξεπεράσει και τα σύνορα. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο και για την αστυνομία να γνωρίζει εάν θα μείνει το δεδομένο μέσα στη χώρα ή αν θα διαβεί και τα σύνορα. Αυτό λοιπόν κάνει δύσκολη τη ζωή τη αστυνομία. Γι' αυτό λέμε ότι θα καλύπτει όλε τι ανταλλαγέ δεδομένων, είτε είναι εθνικέ είτε είναι διεθνικέ, δηλαδή ευρωπαϊκέ. Ευχαριστώ. Ορίστε εσεί. Από τη γερμανική τηλεόραση, ARD τι θα γίνει εάν η όλη διαδικασία για να ξεβρεθεί λύση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου δεν ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές του επόμενου χρόνου. Θα πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, λέτε, ε, γιατί μπορεί να συμφωνήσουν κιόλας να μην αλλάξουν την νομοθεσία, λέτε, αν δεν φτάσουν σε συμφωνία πριν από τις εκλογές, τότε βέβαια θα αποφασίσει το επόμενο κοινοβούλιο. Αν ήδη έχει γίνει ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, μπορεί να αποδεχτεί το επόμενο κοινοβούλιο, που στην επόμενη θητεία δηλαδή, να δεχθεί την ψήφο του του του κοινοβουλίου ή να την απορρίψει. Είναι λοιπόν ανοιχτή. Χωσέ Μανουέλ. Συνήθως το νέο κοινοβούλιο επιβεβαιώνει, ας πούμε, επικυρώνει, λοιπόν, με απόφασή του, το state of play, το που βρίσκεται δηλαδή η διαδικασία. Συνήθως, συνήθως, όπως είπα. Εάν δεν υπάρξει δηλαδή τελική συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογέ, η διαδικασία θα συνεχιστεί. Δηλαδή, το νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές επικυρώνει με απόφασή του την φάση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία από το προηγούμενο, την προηγούμενη θητεία. Όμως, εάν είναι απόλυτα διαφορετική ή πολύ διαφορετική η ε, πλειοψηφία, τότε ίσως να μην θεωρήσει ότι έχει λήξει η διαδικασία και να την ανοίξει. Άλλος κανείς? Μας μένει λίγο χρόνος. Εσείς. Μικρόφωνο παρακαλώ. We have a uni uh, uh, Pathfinder GR. Γιάννης Ριζόπουλος, Pathfinder GR, από την Ελλάδα. Βλέπουμε μια παγκόσμια τάση για ανοιχτά δεδομένα. Έχετε κάνει κάποια σκέψη σχετικά. Από όσο γνωρίζω, η πρόταση της Κομισιόν πάει να καλύψει και τα open data, γιατί και αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Και από τη στιγμή που είναι προσωπικά δεδομένα, σήμερα ισχύει επ' αυτόν ο κανονισμός και θα συνεχίσει να ισχύει. Διότι όπως είπα ο κανονισμός δεν έχει πρόθεση να οπισθοχωρήσει, να πάει πίσω δηλαδή σε σχέση με το σύστημα. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να βελτιώσει το σύστημα, να καταργήσει ή να εξαλείψει τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν ξεπηρήσει τα τελευταία χρόνια, όχι όμως να επανέλθει να δημιουργήσει νέο σύστημα το οποίο θα είναι λιγότερο προστατευτικό, το οποίο θα εξαιρεί διάφορα είδη πληροφοριών κτλ. Εάν είναι προσωπικά δεδομένα, καλύπτονται από, τον, από την οδηγία ή τον κανονισμό. Καλύπτονται επομένω καταρχήν από τον κανονισμό όπως είναι σήμερα και από την οδηγία. Okay. Σύμφωνοι. Ε, επιθυμεί κανείς να καταθέσει άλλη ερώτηση. Θα έχετε βέβαια τη δυνατότητα να ρωτήσετε και τους ίδιους τους ευρωβουλευτές. Αν θέλετε τώρα από εμά τους ε, αξιωματόχους κάποια άλλη πληροφορία. Δεν ξέρω αν το είπαμε. Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα οδηγία και ο κανονισμό από τη στιγμή που θα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, νομίζω η Κομισιόν έχει προτείνει διετία. Ναι, δύο χρόνια. Αυτό δεν το τροποποιούν στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Όχι, μόνο το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να αποφασίσει να ε, κάνει βραχύτερη ή να κάνει μακρότερη την περίοδο αυτή. Πάντως για την ώρα, εφόσον γίνει η τελική έγκριση των δύο αυτών νομοθετημάτων μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νέος εκεί, ε, τέλη 2015-2016. Τώρα μας μένει χρόνος. Ναι. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις τώρα, θα προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ, αλλά πρώτα να σας πω ότι εάν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση email σας όταν γραφτήκατε, όταν καταχωριστήκατε, θα σας στείλουμε τις διάφορες πληροφορίες που είδατε, καθώς και τα PowerPoint και στα ντοσιέ σας. Έχετε και ένα σημείωμα ιστορικού από το Press Service που σας εξηγεί ορισμένα από τα θέματα που τίθεται τώρα. Έχετε και κατάλογο των Ευρωβουλευτών, αν θέλετε να κάνετε κάποιες συνεντεύξεις μαζί τους, εκτός από την αυριανή συζήτηση. Υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο δεν είναι μέσα στο ντοσιέ, αλλά έχει διανεμηθεί εκεί μπροστά, από, σχετικά με τις μελέτες που έχουν κάνει τα διάφορα τμήματα του Κοινοβουλίου. Και αν θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε. Επίσης υπάρχει και ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα μας όπου έχουμε βάλει όλο το υλικό σχετικό με προστασία δεδομένων και με links για τα διάφορα έγγραφα της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Και όταν θα εγκριθούν οι εκθέσεις θα είναι και όλο το σχετικό υλικό. Για την ώρα δεν νομίζω να έχουμε ε, link, δεν υπάρχει... Υπάρχει εδώ τώρα διασύνδεση με το διαδίκτυο. Αν υπάρχει, να σας δείξουμε πού είναι αυτές οι σελίδες την ώρα που θα αλλάζουν τα πρόσωπα του πάνελ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους μου, Ναταλία και Χωσέ Μανουέλ. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις τώρα. Έτσι δεν είναι, μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως. Uh, Ωραία. Περνάμε στο επόμενο πάνελ. Θα το συντονίσει η Κλέρ Νταβενπόχ. Το πρώτο αυτό πάνελ είναι με τον Jean Γκονιέ, που είναι διευθυντής της Privacy Policy Europe, Middle East and Africa της Microsoft και ο Τζέρεμι Τζίμερμαν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της La Quadrature du Net, τετραγωνισμός του δικτύου. Θα βλέπετε και τα Twitter. Οι συμμετέχοντες στα άλλα πάνελ, άμα θέλετε, μπορείτε και εσείς εδώ στο κέντρο να εγκατασταθείτε.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 Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε αυτήν την συζήτηση που πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. ευχαριστώ και όλους όσους μας παρακολουθούν ε, από το διαδίκτυο. Πρόκειται για την ε, προστασία δεδομένων, για τον σχετικό κανονισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται πολύ από τα μέσα ενημέρωση και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και για να είναι πιο ενδιαφέρον το θέμα, να σας πω ότι έχουμε εδώ δύο εμπειρογνώμονες. Πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε για τον ιδιωτικό βίο και το νέφος, το clouding. Έχουμε τον Ζαν Γκονιέ και τον Ζερεμί Τσίμερμαν. Ο πρώτος από τη Microsoft και ο δεύτερος από την εκπρόσωπος ε, της οργάνωσης ο του δικτύου. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από σένα. Σας ευχαριστώ όλους. Δεν υπάρχει μετάφραση, λέει ο μιλητή και θα μιλήσω αγγλικά. Έχει όμως, μπορεί να μιλήσει γαλλικά, μπορεί να μιλήσει γαλλικά. Οι σημειώσει μου όμως είναι στα αγγλικά, λέει ο μιλητής, και γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Θα σας παρουσιάσω την άποψη της Microsoft για ένα θέμα που βέβαια είναι περίπλοκο. Με κάποια απόσταση όμως πρέπει να αντιληφθείτε ότι ζούμε σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Η τελευταία αναθεώρηση για τα θέματα αυτά έγινε το 1995, πριν από 18 χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με την προστασία του ιδιωτικού βίου και τα προσωπικά δεδομένα εδώ και πολλά χρόνια και το 2001 στη Γαλλία και έχω ασχοληθεί πολύ με αυτά τα ζητήματα. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας τα πράγματα προχωράνε γρήγορα. Πολύ σημαντικοί παίκτες, η Google, το Facebook, το Twitter δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια. Δεν ήταν ίδια τα ζητήματα που είχαμε για την προστασία δεδομένων τότε, όπως και τώρα. Δεν ξέρω πώς εξοικειωμένοι είσαστε με την μεταρρύθμιση αυτή. Γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θέλω όμως να κάνω μια νομική αναφορά πριν αρχίσουμε για την προστασία δεδομένων, τον ιδιωτικό βίο. Υπάρχει το άρθρο 8 ενός πολύ σημαντικού κειμένου που είναι Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμολιακών Δικαιωμάτων και καθορίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σαν ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Πολύ βασικό αυτό για όλους μας. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους στον υπόλοιπο κόσμο. Ήμουνα στις Ηνωμένε Πολιτείες πριν από λίγες εβδομάδες και πάντα ε, λέγανε πόσο σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Το άρθρο 8 λοιπόν του Χάρτη Θεμελιωμένων Δικαιωμάτων της Ευρώπης λέει ότι η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει με σωστό τρόπο και αφού προηγουμένως υπάρχει συνένεση. Εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει για το θέμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Και ισχύει συγχρόνως με το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης να μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα. Και γιατί το τονίζω αυτό, διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον της προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Και είμαι πεπισμένος ότι αρχές αυτές είναι πολύ σημαντικές για όλους μας και είναι ακριβώς αυτή η άποψη που έχω για το μέλλον για την προστασία δεδομένων. Εδώ συζητάμε ε, πιο συγκεκριμένα βέβαια για το cloud computing, έτσι. Για το νέφος. Που τι είναι? Είναι ένα σύνολο δεδομένων. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Πάρα πολλοί κόσμος μιλάει για αυτά, για πάρα πολλά δεδομένα, ναι, αλλά τι ακριβώς είναι σήμερα αυτό. Ο καθένας θα έδινε ένα διαφορετικό ορισμό αν ρωτούσαμε. Για μας, για την Microsoft, ήδη εδώ και 15 χρόνια έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δεν είναι για μας κάτι εντελώ καινούριο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι χάρη στις νέες υπηρεσίες που διαθέτουμε, ο καθένας πια αντιλαμβάνεται ότι όπου και να ταξιδεύει, και θέλει να έχει βέβαια τα δεδομένα του οπουδήποτε, ξέρει λοιπόν ότι μπορεί να τα βάλει στον έφος και να τα έχει οπουδήποτε. Για μένα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουν όλοι. Το άλλο που θέλω να συζητήσουμε είναι τις αρχές που για μένα πρέπει να διέπουν τα προσωπικά δεδομένα. Αρχικά ήθελα να μιλήσω μόνο για το clouding, αλλά τώρα σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον για σας να έχετε την άποψη κάποιου από τον κλάδο που έχει δουλέψει στον τομέα αυτό της προστασίας. Ε, ποια είναι η άποψή του λοιπόν για το μέλλον. Η μεταρρύθμιση θα αρχίσει να ισχύει από το 2016. Όμω σε τρία χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά στην προστασία των δεδομένων, στα δεδομένα τα ίδια, γιατί η τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν θα σα δώσω τη δικιά μου οπτική για το μέλλον. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτικό βίο και clouding αν δεν έχουμε υπόψη μα τον όρο διαφάνεια. ο ιδιωτικό βίος, τα ιδιωτικά δεδομένα και η διαφάνεια πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Δεν μπορείτε να έχετε ε, ιδιωτικό βίο χωρίς ε, να βάλετε μαζί το θέμα της διαφάνειας. Η προστασία προσωπικών ε, δεδομένων είναι ένα δικαίωμα. Το βάζετε μπροστά στην πόρτα σας, μην ενοχλείτε, έτσι. Και είναι υποχρέωση από πλευρά των επιχειρήσεων να τηρούν τη διαφάνεια. Εσείς δηλαδή έχετε το δικαίωμα της προστασίας, έχετε το δικαίωμα αυτό και οι άλλοι έχουν την υποχρέωση της διαφάνειας. Για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο δηλαδή. Υπάρχουν προϊόντα της Microsoft προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο που θέλω να συζητήσουμε μαζί σε σχέση με την, τα δεδομένα και το clouding είναι και κάτι άλλο σχετικά πρόσφατα έχει προκύψει και συζητούν οι αρχές και στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και αυτό είναι risk-based approach, δηλαδή η προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο που ελοχεύει. Είναι μια αρχή που έχει συζητηθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, η έκθεση του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρου που αναφέρθηκε στην προστασία δεδομένων συζήτησε πολύ για την χρήση των δεδομένων και για την προσέγγιση αυτή βάση κινδύνου. Εννοείται ότι με το χειρισμό δεδομένων μπορούμε να έχουμε ωφέλη αλλά και ζημιές. Και γι' αυτό πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε την παραδοσιακή προσέγγιση που έχουμε για τη διαχείριση των δεδομένων και να αλλάξουμε. Αντί να επικεντρωνόμαστε μόνο στον έλεγχο των δεδομένων, να επικεντρωνόμαστε και στη χρήση των δεδομένων. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Πώς ο χρήστης ε, μπορεί να ελέγξει καλύτερα το τι γίνεται με τα δεδομένα του. Ο χρήστη του διαδικτύου είναι ο μιλητή προφανώ. Συνεπώ πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή από την προστασία των πολιτών από κάθε κίνδυνο να περάσουμε σε μια άλλη προσέγγιση που να δουλεύει βάση κινδύνου. Δηλαδή ανάλογα με τον κίνδυνο που υπάρχει να μπορούμε να προστατεύσουμε ανάλογα και τα δεδομένα. Δεν θα σας εκπλήσει, αλλά αυτή είναι και η πρόσφατη στάση των κρατών μελών και των αρχών ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτή την προσέγγιση υποστηρίζουν ε, την προσέγγιση προστασία βάση κινδύνου. Γιατί έτσι αποφεύγεται υπερβολικός φόρτος εκεί που δεν χρειάζεται και από την άλλη μεριά μπορούν να μπουν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με τον κίνδυνο. Γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν ελοχεύουν το ίδιο επίπεδο κινδύνου Οπότε υπάρχει διαφορετικός κίνδυνος και άρα μπορεί να υπάρχει και διαφορετική προστασία ανάλογα με αυτόν. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να μπορεί να ελέγξει ο κάθε πολίτης το τι γίνεται με τα δεδομένα του. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας το Fair User Control Model, που συνδέεται άμεσα με τον κόσμο του υπολογιστικού νέφους, του cloud computing. Η διαφάνεια. Η διαφάνεια που σας είπα ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Έχει νόημα, βέβαια, αν επικεντρωνόμαστε στο μέλλον της προστασίας δεδομένων. Κάτι άλλο είναι η μεταβίβαση δεδομένων. Όταν λοιπόν μιλάμε για νέφος και για προστασία δεδομένων, πρέπει να σκεφτούμε πώς μεταφέρονται, πώς μεταβιβάζονται τα δεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόσφατα έγινε μια μελέτη από τον καθηγητή Γέτρο από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα όταν μεταβιβάζονται. Μπορούμε εδώ να σκεφτούμε διάφορα σενάρια να έχουμε προδιαγραφές ίζο, για παράδειγμα. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και μια άλλη προσέγγιση που βασίζεται στη διαφάνεια και αυτό θέλουν οι υπόπτες προστασίας δεδομένων και να σκεφτούμε ένα κόσμο που να βασίζεται στην ε, λογοδοσία. Εγώ είμαι μεγάλος αν με ρωτήσετε τι σημαίνει λογοδοσία, είναι δύσκολο να σας το πω. Πώς είναι, είναι liability, responsibility, πώς μεταφράζεται δηλαδή σε μια άλλη γλώσσα ο όρος accountability, στα αγγλικά λέει ο μιλητής. Σημαίνει προστασία, αξιολόγηση, αλλά πρέπει να πάει με την αναγνώριση, με την αποδοχή Άρα να υπάρχει ένα περιβάλλον που να διέπεται από διαφάνεια. Και μου άρεσε πολύ αυτή η προσέγγιση, γιατί έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να προστατεύσουμε περισσότερο τα δεδομένα και την περίπτωση των δεδομένων που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Α, εσείς τώρα. Γεια σας. Ο Τζέρεμι, είμαι και είμαι hacker. Μην αρχίσετε να τρέχετε για να ξεφύγετε. Είμαι hacker με την πραγματική έννοια της ε, λέξης, δηλαδή είμαι περίεργο, μια περιέργεια για το πώς λειτουργεί η τεχνολογία και έχω και μια πώς πω, φιλοδοξία να την κάνω την τεχνολογία να λειτουργήσει καλύτερα. Hacker δεν πάει να πει ότι χαλάμε τίποτα, θέλουμε να τα φτιάξουμε. Άρχισα με τα τεχνολογικά από πολύ μικρός και πριν από λίγα χρόνια ίδρυσα την, ε, το τετραγωνισμό του δικτύου. Είμαστε πρωτοβουλία πολιτών εδώ και τέσσερα χρόνια. Αναμειγνιόμαστε πολύ σε συζητήσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, παρακολουθούμε τη διαδικασία, φτιάχνουμε tool, εργαλεία για να καταλάβουν οι πολίτες τι συμβαίνει όταν ε, υφίστανται επίθεση οι ελευθερίες μας όχι, σας ευχαριστώ, μην μου δώσετε καφέ. Και εδώ λοιπόν βρίσκομαι σήμερα καθισμένος μπροστά σας να μιλήσω για προστασία δεδομένων. Να είστε βέβαιοι ότι θα προτιμούσα να είμαι αλλού, να είμαι κάπου διακοπές, αλλά νομίζω ότι όντως έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα ως κοινωνία που έχει και βαθιές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Αυτό το cloud τώρα, το σύννεφο αυτό, μου θυμίζει αυτά που λένε και εδώ στην Ευρώπη. Δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ, ανάπτυξη. Δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ, ανάπτυξη. Δηλαδή όλοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα, κανένα δεν ξέρει περί τίνο πρόκειται. Αυτό το cloud είναι απλό πράγμα, δηλαδή δεν είναι και τίποτα το νέο. Cloud θα πει πρώτα-πρώτα virtualization που είναι μια τεχνολογική έννοια όπου αποσυνδέει τα προγράμματα από τους κομπιούτερ, από τους υπολογιστές που τα τρέχουν. Δηλαδή έχεις πολλά κομπιούτερ και ένα πρόγραμμα. Μπορείς να αλλάζεις το σκληρό δίσκο ή τον processor ή οτιδήποτε άλλο, δεν σταματάει τίποτα. Και επίσης virtualization sin outsourcing, δηλαδή να αναθέτεις εξωτερικά κάποια πράγματα. Ότι δηλαδή έχεις εμπιστοσύνη κάποιον άλλο ότι αυτός θα κάνει δουλειά καλά για λογαριασμό σου. Άρα καλό είναι αυτό και για τον λογιστή και για τον διευθυντή IT που δεν θέλει να φορτώνεται το έργο να κάνει όλη τη ε, δουλειά, όλο το computing μόνος του, δώστε τα στο Google, δώστε τα στο Microsoft. Θαυμάσια, μέσα στο σύννεφο να λειτουργήσουν όλα αυτά, πολύ πιο εύκολα. Στη δεκαετία του 80 λέγαμε όλοι, κανείς δεν κάνει λάθος ε, ή κανένας δεν απολύθηκε επειδή διάλεξε να αγοράσει IBM. Τώρα λέμε ότι κανένα δεν απολύεται επειδή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το cloud. Αλλά κανένα δεν ξέρει πώ λειτουργεί αυτό το cloud. Σα είπα ότι εγώ ίδιο είμαι hacker. Τρέχω δίκτυα υπολογιστών για χρόνια. Ξέρω τα MCIP και τα λοιπά, ξέρω πώς να ε, λειτουργήσω ένα σερβερ, αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι για μια στιγμή πώς, ότι γνωρίζω πώς λειτουργεί το ίντερνετ ή πώς λειτουργούν οι υπολογιστές του ίντερνετ. Αυτά είναι πάρα πολύ περίπλοκα πράγματα. Ένας άνθρωπος μόνος του, ένα μυαλό μόνο του δεν πάντα καταλάβει. Αν μπορείτε να καταλάβετε για μια στιγμή τον υπολογιστή, τον επόμενο, την επόμενο δευτερόλεπτο στόσο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να λοιπόν που εδώ είναι κάτι που νομίζω βρίσκεται στην καρδιά του πολιτικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με όλους αυτούς τους κανονισμούς για το διαδίκτυο και τις διαφορετικές τεχνολογίες. Είναι δηλαδή κάτι που κανένα δεν το καταλαβαίνει πραγματικά. Δηλαδή, μεταξύ ημών τώρα, ανοιχτή ερώτηση. Ποιο από εσά ξέρει πού βρίσκονται αποθηκευμένα, physically, πραγματικά δηλαδή, τα email σας. Εσύ ξέρεις, ωραία. Μακάρι να μου πεις και εμένα. ποιο από εσά έχει διαβάσει τα ψηλά γράμματα που λέμε εκτό από τον Τζο εδώ τα ψηλά γράμματα, terms and conditions, ας πούμε δύο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, δηλαδή ας πούμε τα κοινωνικά δίκτυα και το email. Ένας. Μία από αυτές τις υπηρεσίες. Καλώς. Εσείς οι δυο είσαστε οι μόνοι μαζί με τον Ζω. να σας ακούσω να συζητάτε, θα με ενδιαφέρει πολύ. Οι υπηρεσίες, ή μάλλον εταιρείες, όπως το Facebook, ξέρει πότε βλέπετε μια σελίδα που έχει ένα κουμπί like. Αρκεί και να τη δείτε, δεν χρειάζεται καν να το πατήσετε το κουμπί click. Μπορεί να ξέρει και πόση ώρα την είδατε και ότι την είδατε ε, φτάνοντας εκεί από άλλη σελίδα, την χ άλλη σελίδα. Δεν χρειάζεται καμία εξοδότηση για να τα συλλέξει τα δεδομένα αυτά. Η ερώτηση που βάζουμε σήμερα αφού τα δεδομένα έχουν τώρα μεγάλη αξία γιατί πολλούνται τα προφίλ και κάποιοι αποκομίζουν κέρδος από αυτό. Υπάρχει και το ερώτημα των συνεπειών για το μέλλον όταν αποκαλύπτει κανείς όλες αυτές τις προφορίες χωρίς καν να το ξέρει ότι το κάνει. Κανείς εδώ, ούτε οι άνθρωποι του Microsoft, ούτε από την marketing industry μπορούν να σας πούν τι θα γίνουν όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια. Μπορείτε να φανταστείτε 10 χρόνια της ζωής σας στο facebook μπορείτε να φανταστείτε τι θα σημαίνουν αυτά για την τράπεζά σας ή για την interim company που έχετε ή για τον επόμενο εργοδότη σας ή για κάποιον ο οποίος θα ε, αντιπαραταχθεί απέναντί σας σε μια εκλογική εκστρατεία. Άρα πάμε και στοιχηματίζουμε το μέλλον μας ακούγοντας τους ανθρώπους του Microsoft, τον ένα ή τον άλλο που έχουν εμπορικά συμφέροντα να αποκτήσουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα και απλά εμείς τους εμπιστευόμαστε. Α, η διαφάνεια, διαφάνεια φτάνει. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Α, είμαστε ενήλικοι και ούτω καθεξής και όλα θα πάνε καλά. Αυτά λέμε. Εγώ όμως δεν είμαι πεισμένος ότι όλα είναι καλά και ότι όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι η Κομισιόν δούλεψε πολύ για να σχεδιάσει την νομοθεσία. Δεν πάω εδώ να βγω σαν για το λάχ να πω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω στα λίθινα εργαλεία και να γράφουμε μόνο με χαρτί και με μολύβι. Όχι, αυτά είναι βάρβαρα πράγματα του παρελθόντος. Αυτό που λέω είναι ότι αν εξετάσετε την αρχική πρόταση της Κομισιόν θα δείτε ένα κείμενο αρκετά ισορροπημένο, αρκετά προστατευτικό των θεμελιωδών ελευθεριών, με κάποια κενά βέβαια, που νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί, αλλά δεν είναι και τίποτα το επαναστατικό, είναι αρκετά ισχυρό με τον στόχο να επιστρέψει στους πολίτες τον έλεγχο των ζωών τους, του βίου τους, της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν, όπως είναι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, είναι γεμάτη τρύπε, γεμάτη παράθυρα. τέσσερις φιοφορίες στις διάφορες επιτροπές όλες απόλυτα ευθυγραμμισμένες με αυτά που τους ζητούν οι λομπίστες των ε, βιομηχανιών. Όλοι έχουν αποδυναμώσει την αρχική προστασία που προβλέπει η Κομισιόν. Και αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικά και από ότι μέλλον είναι αυτό το μαζικό λόμπι των εταιριών που στην ουσία υπαγορεύει τι θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία δεδομένων. Που στο κάτω τη γραφή κανένα δεν ξέρει τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε, ε, βλέπω εγώ ένα έντονο δημοκρατικό πρόβλημα. Πώς να πει κανείς τώρα bullshit εδώ στο ε, ανοιχτό μικρόφωνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα μόλις το είπες, του λέει πλανήτη. Αυτά θα σας πούνε. Α, κάποιος θα σας πει εδώ ψευδόνυμα, ψευδόνυμα δεδομένα. Α, ωραία, ας βάλουμε ψευδόνυμα, πολύ ωραία, ας το κάνουμε αυτό αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι 90% των προφίλ των ψευδόνυμων μπορούν να ανακληθούν. Κάποιος που δουλεύει πάνω σε μια βάση δεδομένων, αυτό που κάνουν κάθε μέρα είναι να διασταυρώνουν δεδομένα για να κάνουν recall information. Είναι τρίχε αυτά λοιπόν. Είναι απάτε. Δεν σημαίνουν απολύτω τίποτα. Όμω το κοινοβούλιο πάει να το ψηφίσει. Ίσως και να το ψηφίσει. Άρα το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται για να σα καταστρέψουν την προσωπική σφαίρα. Σας είπα πριν η γλώσσα της Ευρώπης που είναι jobs, jobs, growth, growth. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, αυτό που θα έκανε νομοθέτη θα ήταν να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια αγορά διαδικτύου ευρωπαϊκή βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους online operators. Αν μπορούσαμε να τους βάλουμε, να βάλουμε τέτοιες συνθήκες που να τους λέμε ότι μπορείτε να τους εμπιστεύεστε γιατί είμαστε εδώ Ευρώπη, νομίζω τότε ότι θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό απέναντι στις ΗΠΑ και πολύ περισσότερες δουλειές από ό,τι έχουμε σήμερα. Τέλος, ένα σύντομο συμπέρασμα. Το θέμα αυτό είναι πολιτικό, καθαρά. Έρχονται οι εκλογές. Βλέπετε, είδατε τον κόσμο να κατεβαίνει στους δρόμους για το άκτα. Σε 300 πόλεις και στις 27 χώρες μέλη να μιλούν για την πολυμερή διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Αυτό όμως εδώ είναι πολύ πιο περίπλοκο, αλλά είναι το ίδιο πολιτικό όπως και το άκτα. Και ελπίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες θα σας το αποδείξουν. Ευχαριστώ, Τζέρεμι. Ευχαριστώ. Τις ίδιες ανησυχίες έχεις και εσύ, Τζέρεμι. Μετά από 10 χρόνια δηλαδή στο Facebook. Μα είπα και πριν και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και βλέπω αυτά τα οποία μας λέει τώρα ο Τζέρεμι. Γι' αυτό και τόνισα τη διαφάνεια πριν. Αν υπάρχει μία λέξη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, είναι εμπιστοσύνη. Αλλά την εμπιστοσύνη την κερδίζει κανείς. Στην αρχή μιας σχέσης δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, χτίζεται. Δεν είναι λάθος η ανησυχία. Συμφωνώ ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη και αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίζεται μέρα τη μέρα. Από την Microsoft θα το προσπαθήσουμε γιατί το ξέρουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο του δικτύου. Για κάθε λοιπόν cloud θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και να μπορεί έτσι ο κάθε πολίτης να βλέπει πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα. Έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και θα αναπτυχθεί, γιατί αλλιώ δεν θα κερδιθεί αυτή η επιστήμη που ε, πρέπει να υπάρχει. Και θα έλεγα και άλλες εταιρείε πρέπει να κάνουν το ίδιο. Ρώτησες πριν πού τοποθετούνται τα δεδομένα. Εγώ ξέρω για την Microsoft. Το Hotmail που μπορεί να έχετε και ελπίζω πολλοί από εσά να έχετε λογαριασμούς Hotmail αποθηκεύονται στην Ευρώπη. Αν είσαστε Ευρωπαίος πολίτης στην Ιρλανδία ή στις κάτω χώρες. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε δεσμευτεί για αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε πού βρίσκονται αυτά τα δεδομένα. Εμείς ξέρουμε τα δικά μας, αν είσαστε Ευρωπαίος πολίτης, είναι στην Ευρώπη. Θέλω επίσης να τονίσω και κάτι ακόμα. Και πάλι για τη Microsoft βέβαια μιλάω. Ε ότι καθημερινά, καθημερινός διευθυντής ε, που είμαι για την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη, Αφρική κτλ. Από την αρχή, εξ αρχής, δουλεύουμε με αρχές για την προστασία δεδομένων. Εννοείται ότι δουλεύουμε με ρυθμιστές. Είναι φυσιολογικό. Εμείς στη Microsoft προστατεύουμε καλύτερα τα δεδομένα όταν μεταβιβάζονται ανά τον κόσμο. Και αυτό γιατί έχουμε συζητήσει με τους επόπτες. Αναφέρθηκες και στην πιστοποίηση. Μα κοίταξε και τι κάνει η Microsoft. Εγώ είμαι υπέρ και συμφωνώ μαζί σας. Από τη στιγμή που υπάρχει από τον Ευρωπαίο επόπτη μία label, να ξέρετε ότι θα υπάρχει, αλλά δεν έχει καμία αξία αν δεν συνοδεύεται με επιβολή. Έχουμε και σήμερα ε, τις περισσότερες φορές κάποιον κώδικα θεοντολογίας. Οι διάφορες οδηγίες που υπάρχουν δεν χρησιμοποιούνται γιατί, γιατί υπάρχουν κάποια κενά και τελικά δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή Καλό είναι να υπάρχει επιστοποίηση, αλλά πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την επιβολή, με την εφαρμογή. Δεν ξέρω πώς, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει και αυτό το στοιχείο της υποχρεωτικής εφαρμογής ή επιβολής. Και κάτι ακόμα έχω να πω. Ο, ο επόπτης δεδομένων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν ελέγχουμε τα δεδομένα μας όταν δεν τα γνωρίζουμε. Τα cookies. Τι είναι τα cookies. Υπάρχουν cookies που είναι ενδιαφέροντα, αλλά που είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια ενημέρωση, κατάρτιση για αυτά. Αν δεν τα καταλάβουμε τι είναι τα δεδομένα μας, δεν μπορούμε και να τα προστατεύσουμε σε πολλές χώρες γίνεται αυτή η ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο έλεγχος δεδομένων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ερωτήσεις. Έχουμε 20 λεπτά για ερωτήσεις. Οπότε παρακαλώ, ποιος ε, έχει ερώτηση. Παρακαλώ. Εσείς. Ναι. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο αν πάω στη Microsoft και ρωτήσω, για μένα, τι δεδομένα έχετε, θα μου απαντήσουν. Ευχαριστώ. Ναι. Απάντηση. Ναι. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ξέρετε εσείς τι δεδομένα βάζετε στο διαδίκτυο. Γιατί αυτό είναι το παράδοξο του ιδιωτικού βίου. Γιατί όλοι μας θέλουμε να βάλουμε τη ζωή μας στο διαδίκτυο και μετά διαμαρτυρόμαστε ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Βεβαίως και θα σας απαντήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να ξέρετε εσείς τι δεδομένα βάζετε στο διαδίκτυο. Εγώ προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός με τα δικά μου δεδομένα ή των παιδιών μου. Να μην βάζει κανείς δηλαδή στο διαδίκτυο δεδομένα για το οποίο θα μετανιώσει αργότερα. Να απαντήσω κι εγώ κάτι σε αυτό λέει ο κύριος Τζίμερμαν. Ένας φοιτητής νομικής στην Αυστρία πέρασε δύο χρόνια να δίνει αγώνα με το Facebook γιατί για να μπορέσει να ασκήσει τα δικά του δικαιώματα ως Ευρωπαίος πολίτης για να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αυτός είχε βάλει στο Facebook. Δύο χρόνια του πήρε η διαδρομή ανάμεσα στα διάφορα ένδικα και μη μέσα. Ξέρετε ότι η έδρα είναι στη, στο Δουβλίνο. Τελικά πήρε ένα DVD 900 MB για τα δεδομένα που είχε η Facebook τα δικά του. Ακόμα και για όλα εκείνα στο οποίο είχε κάνει delete, ακόμα και για ό,τι είχε διαγράψει από το διαδίκτυο, υπήρχαν στο Facebook. Τα είχε η Facebook. Τέτοιου είδους συμπεριφορά λοιπόν είναι απαράδεκτη δεν πρέπει να υπάρχει με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το θέμα της συμμόρφωσης ε, με τις διάφορες νομολογίες κτλ. δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά σίγουρα περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον να κάνει αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή. Τουλάχιστον. Και όχι να το κάνει σουρωτήρι ανοίγοντας τρύπες δεξιά και αριστερά. Θέλω επίση να σας ρωτήσω, σε ποιο κομπιούτερ, σε ποιο ρακ, σε ποιο κέντρο δεδομένων της Ιρλανδίας ή των κάτω χωρών είναι τα δεδομένα του δικού σας λογαριασμού email. Δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε. Πάντως η τρέχουσα κατάσταση, όταν βλέπετε Facebook, Yahoo και τα λοιπά, οι εισηγητέ για την προστασία των καταναλωτών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνουν copy-paste από το Google, είπαμε κι αλλού. Ε, τελικά τι κάνουν, αντιγράφουν αυτά που θέλει η βιομηχανία. Πώς θα μας πούνε λοιπόν ότι είναι καλό για μας. Άλλη ερώτηση. Εσείς πρώτος ήσασταν εκεί με τα λευκά. Τσέχος δημοσιογράφος γιατί δεν είναι απλώς δυνατό να δοθεί σε κάθε χρήστη, σε κάθε καταναλωτή, απλά η τεχνική δυνατότητα να πει δεν θέλω τα δεδομένα μου να τα επεξεργαστεί κανένας ούτε να χρειαστεί κανένας. Γιατί για παράδειγμα Microsoft στα Windows δεν βάζει ένα τέτοιο μηχανισμό και επίσης και σε, και σε άλλα λογισμικά. Γιατί δεν είναι δυνατό αυτό. Καλή ερώτησή σας. Με εκπλήσει, αστείευομαι, που θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Γκονή, αλλά αυτό που έχει σημασία πρώτα-πρώτα είναι που, να γνωρίζετε πού τα βάζετε τα δεδομένα σας είμαι hacker όπως σας είπα και είχα την τύχη να μάθω για υπολογιστές από τότε που ήμουν μικρό παιδάκι. Ξέρω, πρέπει να ε, χρησιμοποιείτε τον δικό σας σερβερ, να κάνετε encrypt τα δεδομένα σας. Υπάρχουν και μερικές, μερικά μέτρα που μπορεί να πάρει κανένας, ώστε να μην μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να αντιληφθεί ο καθένας πού βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στο privacy, intimacy ένας κύκλος εμπιστοσύνης, κάποιου δηλαδή στου οποίου έχετε εμπιστοσύνη και με αυτούς θέλετε να μοιραστείτε κάποιο φορεί, και τι είναι δημόσιο, τι είναι public. Έχετε εταιρείε όπως Facebook, Google και άλλα που το ίδιο το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στο να θολώνουν τα όρια αυτά. Να σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσεί βρίσκεστε μεν μέσα σε ένα κύκλο εμπιστοσύνη όταν μοιράζεστε πληροφορίε με του φίλου σα στο Facebook Α, είναι όμως αυτός ο κύκλος εμπιστοσύνη συν όλοι οι άλλοι που είναι στο facebook. Ναι, θα χρειαστούμε λοιπόν κάποια εκπαίδευση για τα παιδιά, για τους ε, νέους όταν θέλουν να είναι star και να έχουν πολλούς φίλους αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε βέβαια ενάντια σε αυτές τις εταιρείε, όταν αυτές οι εταιρείε συνεχίζουν όπω είπα να θολώνουν τα νερά τα όρια δηλαδή ανάμεσα στην privacy και στην publicity από την άλλη μεριά. Το ερώτηση σας Α, ναι, ναι. Ναι, η συνένεση του χρήστη δηλαδή να μπορεί ο ίδιο να αποφασίζει τι θέλει να βάλει και τι δεν θέλει ως προσωπικά δεδομένα. Σε κάποιον, όχι ακριβώς, η ερώτησή μου είναι γιατί δεν υπάρχει ένα απλός τρόπος με τον οποίο ο χρήστη να μπορεί να αποφασίσει πώς μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του. Το κατάλαβα και εκεί σας απαντούσα. Είναι από τα κέρια σημεία που συζητούνται τώρα στις συμβαστικές τροπολογίες στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Από τα κέρια θέματα λοιπόν το ζήτημα της συνένεσης. Ποια απέτηση επιβάλλουμε στις εταιρείες αυτές για να ζητήσουν την συνένεση των χρηστών. Αν βάλουμε αυστηρές απαιτήσει, θα μας πούν Είχαμε μέχρι τώρα όλε τι εικόνε, τι φωτογραφίε σα. Τώρα θέλουμε να βάλουμε και τα γεωγραφικά σα δεδομένα. Α, ή έχουμε τα γεωγραφικά σα δεδομένα, θέλουμε ακόμα και το Α ή το Β. Ναι, όχι. Αν δεν του βάλουμε κάποιο περιορισμό να είναι πάρα πολύ ακριβεί σε ό,τι αφορά τη συνένεση που θα πρέπει να λάβουν από το χρήστη, τότε έχουν οικονομικό κίνητρο να κάνουν τα άλλα. στο τέλος των 80 σελίδων ψηλά γράμματα που δεν έχετε διαβάσει, το λέει. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση, απαντά ο Τσέχος δημοσιογράφος, διότι όλοι έχουν την ερώτηση αυτή αν τα δεδομένα τους μπορούν να τύχουν επεξεργασίας ή όχι. Είτε συμφωνείς λοιπόν και άρα μπορεί να χρησιμοποιήσεις το λογισμικό, είτε δεν συμφωνείς και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Αυτό είναι γελίο. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο που να μπορώ να μπω και να πω όχι, δεν θέλω δεδομένα αυτή α πούμε τη περίοδου ή από αυτό τον υπολογιστή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πουθενά άλλου. Και εκεί, stop, τέλο. Αυτό είναι και το νόημα τη απαντήσεώ μου αντί να έχουν μια σύμβαση 80 σελίδων που σας δίνουν να διαβάσετε όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό και που μπορείτε είτε να τη δεχτείτε να τα απορρίψετε στο σύνολό της, να είναι σε μικρότερες, πιο κατανοητές ενότητες που αν απορρίψετε τη μία να μην σας αναγκάσει να απαρατηθείτε από τη χρήση ολόκληρου του λογισμικού αλλά αυτό μπορεί να επιβληθεί μόνο από τον νομοθέτη. Δεν μπορείτε να αναμένετε από τους ε, κατασκευαστές. Τζον, θέλετε να ασχολείστε. Ναι, βέβαια. Πρώτα ευχαριστώ για την ερώτηση σας. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που θέσατε την ερώτηση. Να έρθετε να δείτε το κέντρο μας, γιατί αυτά δουλεύουμε τώρα. Και θέλω να σας εξηγήσω, γιατί νομίζω ότι έχετε δίκιο. Μιλήσαμε για τη διαφάνεια και ο έλεγχος από το χρήστη είναι το κλειδί. Πολύ σωστό από την αρχή ως χρήστης να μπορείτε να χειριστείτε τα δεδομένα σας. Να μπορείτε να πείτε δεν θέλω αυτό, θέλω αυτό. Αυτό δεν μου κάνει, εκείνο μου κάνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ε, δουλεύουμε τώρα στο Windows 8 και στο Windows Blue που θα είναι το επόμενο. Είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβει μια επιχείρηση Αυτό να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Do not track είναι μια δυνατότητα που μπαίνει by default στο Windows 8 για να απορρίπτεται η στοχευμένη διαφήμιση. Γιατί αυτό ακριβώς ενοχλεί πολλούς και παραπονούνται. Αυτό για πολλούς λόγους είναι δύσκολο να επιτευχθεί η συνένεση με την υπόλοιπη βιομηχανία, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί η Microsoft σήμερα είναι η μόνη επιχείρηση που το κάνει. Καλό είναι να γίνεται συζήτηση, ακόμα καλύτερα να έχουμε συγκεκριμένε αποδείξεις. Δεν μπορώ να σας πω τώρα περισσότερα παρά αυτό μόνο το συγκεκριμένο. Καμιά ερώτηση ακόμα εκεί πίσω εσείς. για τον κύριο Γκόνη. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μιλήσατε για διαφάνεια και για τη δημιουργία εμπιστοσύνη. Επομένως, εάν υπάρχουν ε, παραβιάσεις θα τις ε, καθαστήσετε ε, δημόσιε στο μέλλον. Βλέπω και την οδηγία. Γίνεται συζήτηση σήμερα για το data breach και ιδίω για την κοινοποίηση στι 24 ώρες. Αλλά αν υπάρχει ο κανόνας θα ακολουθούμε τον κανόνα. Αλλά όπως όλοι είμαστε διαφανεί. από τη στιγμή που υπάρχει notification που να γνωρίζουμε την καθιστούμε γνωστή στην τοπική αρχή. Να κάνω μια μικρή προστίκη. Ή έχετε και άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Αυτό είναι επίσης πολύ κέριο θέμα της νομοθεσίας και πάει να αποδυναμωθεί κάτω από την πίεση της βιομηχανίας. Δεν θέλουν να αποκαλύπτουν στους χρήστες τους data breach. Α, γιατί τότε σημαίνει ότι δεν έχουν, ε, δεν έχουν ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Γνωρίζετε περιπτώσεις με χιλιάδες ε, ε, tracks και records κτλ. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε μάλλον στοιχεία ότι τέτοιες εταιρείες δεν χρησιμοποιούν την, την πιο σύγχρονη τεχνολογία για την προστασία των δεδομένων. Και τώρα πάει το Κοινοβούλιο να μειώσει τις υποχρεώσεις που ε, επιβάλλονται σε εταιρείες αυτές να μας ειδοποιούν για data breach, για παραβιάσεις το, της ασφάλειας των δεδομένων. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ οργανώσεις Ευρωπαίων καταναλωτών. Λίγα λόγια για την συνένεση, η συγκατάθεση. Πιστεύω ότι πρέπει όντως να υπάρχει δυνατότητα του καταναλωτού να δίνει τη συγκατάθεσή του που να είναι ο νομικός λόγος για την συλλογή των δεδομένων. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο. Αναφέρθηκαν πριν οι ε, διατάξει τη ε, οδηγία του 95 που είναι πολύ σημαντικές και η συγκατάθεση πρέπει να είναι σκόπιμη. Δηλαδή πρέπει η συγκατάθεση να, να ε, συνοδεύεται από την συμμόρφωση του ελεγκτή. Άρα να συλλέγω τα δεδομένα σας για συγκεκριμένους σκοπούς, όχι για ό,τι θέλει ο ελεγκτής. Επίσης η κατάθεση δεν σημαίνει τίποτα χωρίς διαφάνεια. Χωρίς μια καλή πολιτική διαφάνειας. Δεν χρειάζεται να σας πω Δεν πιστεύω κανένα να έχει διαβάσει από εσά την privacy policy των μεγάλων εταιριών. Γιατί για να το κάνετε αυτό θα σα χρειαστούν χρόνια. Μου φαίνεται ότι υπάρχει και άλλη ερώτηση. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη ερώτηση. Άλλος κανείς. Για αυτήν την διαφάνεια, λέει ο Τζέρεμι. Αυτό είναι από αυτές τις λέξεις συνθήματα, job, jobs, growth, growth, που την χρησιμοποιούν και τη χρησιμοποιεί η βιομηχανία διαρκώς όταν θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε ρύθμιση και οποιαδήποτε, οποιοδήποτε περιορισμό. Βλέπουμε την ίδια τάση και στην συζήτηση για την ουδετερότητα του διαδικτύου και το ίδιο και στο πακέτο τηλεπικοινωνιών 2009-10 ότι η διαφάνεια φτάνει από τη στιγμή που μέσα στη σύμβασή σας κάποιος λέει πώς γίνεται η πρόσβαση στη, στο δίκτυο ε, μπορείτε να αλλάξετε operator ναι. αλλά αυτό χρησιμοποιείται συχνά και σαν προπέτασμα καπνού και σαν εναλλακτική επιλογή στην ρύθμιση, στη regulation της ε, βιομηχανίας. Ναι, ο Τζο. Θέλω και εγώ να προσθέσω κάτι στην απάντηση που έδωσες. Πριν από μερικά χρόνια, όταν για το διαμέρισμά μου ε, κατέληγα σε μια συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία, ήταν σε χαρτί και έλεγε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για να τα χρησιμοποιήσουν για διαφήμιση. Τώρα όμως, χάρη στη νέα τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε να κάνουμε πριν, λιγότερα, μπορούμε να κάνουμε λιγότερα από όσα μπορούσαμε να κάνουμε τότε με το χαρτί. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πρέπει να λένε ποια δεδομένα είναι υποχρεωτικά και ποια δεν είναι υποχρεωτικά ποια πρέπει να δίνετε και ποια μπορείτε να μην δίνετε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αντιπρόσωποι μας, αυτοί για τους οποίους θα ψηφίσουμε του χρόνου, έχουν υποβάλει τροπολογίες με τις οποίες θέλουν να διαγραφεί αυτό. Και ξέρω ότι μας βλέπουν και από βίντεο. Δεν είναι δυνατόν να πάμε προς τα πίσω, να έχουμε πιστοχώρηση δηλαδή. Καλώς ήταν η τελευταία παρέμβαση. Κοιτάξτε, μάλλον τώρα η τελευταία ερώτηση. Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται λιγότερο το νέφος από ότι αλλού. Γιατί υπάρχει λιγότερη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη προς τις εταιρείε που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που βρίσκονται εκεί ή όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρώπη βρίσκεται τόσο πιο πίσω από τον αντίστοιχο αμερικανικό κλάδο. Ίσως είναι θέμα ανατροπίας. Στην Ευρώπη έχουμε πολλά εθνικά υπολογιστικά νέφη, το γαλλικό, το γερμανικό κτλ. Όμως τα πράγματα πάνε γρήγορα. Αν δείτε τις τοποθετήσεις των διαφόρων κυβερνήσεων, ε, όλες έχουν αποφασίσει να το χρησιμοποιούν. Νομίζω δηλαδή ότι μειώνεται η διαφορά μας με τις ΗΠΑ. Τσίμερμα, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Αν είχαμε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είχαμε μια ενιαία πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι, ίσως και οι πολίτες να συμμετείχαν περισσότερο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να μένουν τα διάφορα λόμπι στα οποία συντάσσουν τελικά την νομοθεσία. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ περισσότερους επικεφαλής ε, ελεύθερων ε, προγραμμάτων από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στο free software. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτούμε τέτοια προγράμματα τα οποία γίνονται στα πανεπιστήμια μας, ε, στα εργαστήρια, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα μπορούσε τέτοιο να χρησιμοποιηθεί και για το υπολογιστικό νέφος. Τελικά, ίσως χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να δουλεύει για τους πολίτες και όχι για τα λόμπις και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Right, so Καλώς, περνάμε λοιπόν στην επόμενη. Περνάμε στην επόμενη συζήτηση που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις του profiling. Έχω δεξιά μου τον κύριο Μακνή και αριστερά μου τον κύριο Ζορμπά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο. Παρακαλώ. Θα αρχίζω από εσάς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. πάει πάση περιπτώσει, Κλέρ, κοιτάω γύρω μου δεν βλέπω πολλέ γραβάτε ούτε κι εγώ. Α, να μία. Να, κι άλλη μία γραβάτα. Να, ε, από οικονομικέ εφημερίδες σίγουρα. Γνωστό αυτό. Α, και αυτό είναι profiling. Προσπαθούμε να καταλάβουμε δηλαδή αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, να δω ποιο είναι το κροτήριό μου, κάνω κάποιες υποθέσεις ο πρώτος εδώ με την κραβάτα δεν είναι καν δημοσιογράφο. Τέλο πάντων, αυτό είναι το profiling. Η συγκέντρωση δηλαδή γνωρισμάτων, χαρακτηριστικών του ατόμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλαβαίνω γιατί σκέφτηκε ότι έπρεπε να αλλάξει το άρθρο 15 στην ε, σημερινή οδηγία. Το έκανε πάντως με κάποιο τρόπο ώστε να διευρυνθεί το εύρος εφαρμογής της. Και τώρα συμπεριλαμβάνει και δραστηριότητες οι οποίες είναι πολλές και διάφορες. Κανονικά περιμένεις το FBI, το MI6, το MI5 να κάνουν το profiling και τελικά διαπιστώνεις ότι το κάνουν οι εφημερίδες, στι οποίες δουλεύετε, το κάνουν τα τηλεοπτικά κανάλια στα οποία δουλεύετε, ραδιοφωνική σταθμή. Και γιατί? Γιατί έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε αυτόματη επεξεργασία δεδομένων τελικά μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά σας ή στις νομικές επιπτώσεις ε, μπορεί να είναι αυτό το profiling βλέπετε διαφημίσεις online. Ε, η διαφήμιση έχει σκοπό να αλλάξει τη συμπεριφορά σας. Χρειάζονται αυτά που προτείνει ο νόμος και ποια είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα ο νόμος θέλει απλοποίηση, ναι, αλλά βασικά τι λέει ο νόμος. Λέει ότι αν δεν επιτρέπεται ρητά από τον νόμο το profiling, τότε απαγορεύεται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διάταξη ρητά στην εθνική νομοθεσία για να το κάνετε. Αυτός είναι ένας περιορισμός από τον νόμο. Ο δεύτερος είναι ότι χρειάζεται συγκατάθεση της άλλης πλευράς και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Για πολλές δραστηριότητες έχει νόημα αυτό, αλλά για άλλες δεν έχει νόημα. Και έτσι ερχόμαστε σε αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για το θέμα της συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση είναι κάτι που λειτουργεί σαν προειδοποίηση στη σημερινή νοοτροπία. Η ρητή συγκατάθεση σήμερα απαιτείται μόνο για την διαδικασία ευαίσθητων δεδομένων. Και σωστά. Γιατί θέλουμε κανείς να σκεφτεί δυο φορές πριν μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο κάτι που θεωρεί ευαίσθητο για την περίπτωσή του. Η τωρινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν ζητάει οι χρήστες να δίνουν τη συγκατάθεσή τους ρητά για οποιοδήποτε δεδομένο που τους αφορά. Η σελίδα σας, για παράδειγμα. news.com Τι κάνει αυτό το site, προσπαθεί να καταλάβει ποια κομμάτια website είναι καλά για το χρήστη, ποια ανοιχνεύουν το τι χαρακτηριστικά έχει ο χρήστη, ή αυτό μπορεί να βοηθάει μερικέ φορέ τον δημοσιογράφο, γιατί έτσι μαθαίνει πόσοι έχουν διαβάσει το άρθρο του. Είναι κακό αυτό. Κανεί όμω δεν θα πάει πίσω και θα του πει του χρήστη Α, είδαμε τι έχει κάνει. Όχι. Πρόκειται για ε, συσσόρευση δεδομένων για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του κόσμου, τις αντιδράσεις του κόσμου. Οι εφημερίδες, για παράδειγμα, θέλουν να ξέρουν τι ποσοστό του πληθυσμού τις διαβάζει. Ώστε να ξέρουν το 15% του πληθυσμού. Και αν μπουν περισσότερο σε βάθος θα δούνε ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, είναι αυτοί που είναι διευθυντές επιχειρήσεων και έτσι ξέρουν ανάλογα πόσο καλή δουλειά κάνουν ή όχι. Για παράδειγμα, Financial Times. Τώρα, για τα δεδομένα αυτά, οι δικέ μου επιχειρήσεις που κάνουν τέτοια αναλυτική δουλειά, λένε στους πελάτες μας ότι δεν πρέπει να κρατάνε τα δεδομένα πολύ καιρό, γιατί δεν έχει νόημα. Όλοι λένε ότι είναι πολύ φτηνό. Ναι, είναι φτηνό πιο φθηνό στο παρελθόν το να συγκεντρώνει κανεί δεδομένα και να τα αποθηκεύει, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται πολλά χρήματα για να τα αποθηκεύει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και συμβολεύουμε του πελάτες μας να μην το κάνουν για πολύ καιρό. Τώρα τα θέματα ε, πιστοτικά, ασφαλίσεων, σχολεία. Ποιος είναι ο καλύτερος της τάξης, για παράδειγμα, και τέτοια ο νόμος πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικός και δεν αναγνωρίζει ότι κάποια δεδομένα αποθηκεύονται ο κόσμος δεν θέλει να δίνει τη συγκατάθεσή του για αυτά. Για παράδειγμα, έχω κάποιους που δημοσιεύουν ε, κάποιες ειδήσει και του λένε «Εγώ δεν θέλω οι χρήστες να μου δίνουν λεπτομέρειες, δεν θέλω να ξέρω ποιοι είναι». Κανένας δεν θα μου έχει εμπιστοσύνη αν πάω και τον ρωτήσω στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Ιράν να μου δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του. Δεν θέλουν. Μερικές φορές δηλαδή ο κόσμος δεν το θέλει. Συνεπώς, αυτά βέβαια σας τα λέω πολύ περιληπτικά για να κάνετε και ερωτήσεις, να μην φάω όλο το χρόνο. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στη σημερινή συζήτηση. Ο Τζο, αναμφίβολα, θα πει και αυτός περισσότερα πράγματα για το profiling. Υπέροχο δεν είναι αυτό ο Κίμων, Σε κάνει και αισθάνεσαι τόσο άνετα όλοι, τόσο ευτυχισμένοι. Τώρα, κοιτάξτε, σύντομη εισαγωγή. Εκπροσωπώ την Άντρη, οργάνωση σε όλη την Ευρώπη. Όσοι δεν ακούσατε τη σχετική εισαγωγή πριν, έχουμε και έναν οδηγό για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Org, κάθετος, papers καθώς και το Naked Citizens.eu. Όταν μιλούσε ο Ζαν προηγουμένως για διαφάνεια, μου θύμισε μια συνέντευξη που είχα δει με έναν συντηρητικό πολιτικό που έχει αποχωρήσει από την πολιτική ζωή και πώς ήταν να περάσει από τον επιχειρηματικό κόσμο στον πολιτικό. Είναι θαυμάσιος επιχειρηματικός μας, είπε, διότι εκεί σε μαχαιρώνουν από μπροστά τουλάχιστον. Η διαφάνεια λοιπόν έχει ίσως ενδιαφέρον για την big business και η Microsoft αυτή είναι big business. Θέλουν διαφάνεια βασισμένη σε risk-based approach, contact-based approach και technology-based approach καθώς και σε balance of rights based approach. Εάν είσαστε καλός δικηγόρος και δουλεύετε για μεγάλη εταιρεία όπως ο Jean, αυτό είναι απόλυτα λογικό. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, είναι διαφάνεια με την έννοια ότι σε μαχαιρώνουν από μπρο. Διότι δεν λέει βέβαια στον κόσμο τι γίνεται, δεν λέει στου πολίτε τι συμβαίνει. Οι αγορέ δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρί εμπιστοσύνη. Αυτό τουλάχιστον διδαχτήκαμε από την τραπεζική κρίση. Εάν τώρα η Ευρώπη θέλει να υποφεληθεί και αν θέλει να προστατεύονται οι πολίτες, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τη χρειαζόμαστε και εμεί, τη χρειάζεται και η ε, επιχειρήσεις. Ωστόσο υπάρχει βαθιά κρίση εμπιστοσύνης από των πολιτών για το πώς επεξεργάζονται οι εταιρείε τα δεδομένα τους. Μόνο 22% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι ελέγχουν τα δεδομένα τους και μόνο 26% εμπιστεύονται τις online εταιρείε. Άρα, ποια είναι η αντίδραση τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης. Κρίση εμπιστοσύνης που πρέπει να διορθωθεί για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Πρότειναν οι ευρωβουλευτέ. Θα σα διαβάσω τροπολογίε μονάχα για ένα άρθρο. Προτείνουν να επιτρέπετε στις επιχειρήσεις να ε, επεξεργάζουν τα στοιχεία σας χωρίς πρώτερη συγκατάθεση, να τα περνούν σε άλλες εταιρείες χωρίς πρώτερη συγκατάθεση, να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για τρόπους που δεν είναι συμβατοί για λόγους που δεν συμβατεί με αυτούς που είπατε στην αρχή, να σας κρατούν, να παρακρατούν πληροφορίες σχετικά με παράπονα, να τους επιτρέπετε να μην σας λένε αν θα εξαγάγουν τα δεδομένα σας εκτός Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παρακρατούν πληροφορίες για το πόσο χρόνο θα διατηρούν τα αποθηκεύουν τα δεδομένα σας. Αυτές είναι οι προτινόμενες λύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κρίση εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η προτινόμενη λύση από τη βιομηχανία σε περίοδους κρίσεως. Σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων και τη σχετική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις στην ουσία ζητάν αρκετό σκηνή για να μπορέσει να κρεμαστεί από μόνη της και οι βουλευτές αυτό συζητούν πόσο σκηνή θα τους δώσουν. Profiling τώρα. Εμείς το profiling το βλέπουμε λίγο διαφορετικά από τον Κίμωνα Ζόρμπα. Όπως είπε και ο Τζέρεμι πριν, το profiling αλλάζει. Το, το ποσό δεδομένων που συλλέγεται και που ανταλλάσσεται μεταξύ βάσεων δεδομένων αλλάζει. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτς πριν από λίγες εβδομάδες μόνο, που εμένα πραγματικά με σόκα. Εγώ θεωρούσα ότι είμαι απεσιόδοξο, αλλά τελικά αποδεικνύομαι αισιόδοξο σε σύγκριση με αυτά που λέει η μελέτη του Κέμπριτς πήραν ένα σχετικά μικρό ποσοστό δεδομένων από τη δραστηριότητα του Facebook και μπόρεσαν να καταλήξουν με εύλογη πιθανότητα ακρίβειας στη βάση των κλικ όταν ένας καταναλώνει τσιγάρα ε, ποτά μπορούν να γνωρίζουν τις ε, σεξουαλικές, σεξουαλικές προτιμήσεις εσείς δεν γνωρίζετε, ούτε εγώ θα γνώριζα αν χρησιμοποιούσα το Facebook. Τι σας κάνει να πατήσετε το κουμπί like. Αλλά το Facebook στη βάση των αναλύσεών του εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων δεδομένων γνωρίζει τι σημαίνει αυτό το like που πατάτε. Τι προτείνει γι' αυτό τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι πρότειναν δηλαδή τα λόμπι ώστε να τα προωθήσει ως τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ακούσαμε πριν, δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει ρητή συγκατάθεση για το profiling. Θα είναι δυνατό λοιπόν τα δεδομένα να διαβιβάζονται σε τρίτους. Θα είναι δυνατόν οι χώρες μέλη θα μπορούν οι χώρες μέλη να έχουν το δικαίωμα να αυτοεξαιρούνται από ολόκληρη την ισχύ του άρθρου για το profiling. Η δραστηριότητα profiling που διενεργείται θα σημαίνει ότι μπορούν τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με την αρχική συλλογή τους. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Στην ουσία σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη υπονόμευση της εμπιστοσύνης. Και η εισβολή στην προσωπική σφαίρα του καθενό, αρχίζει και γίνεται τώρα εμφανής, όπως είδαμε και από τη μελέτη που σας ανέφερα πριν του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ προ λίγων εβδομάδων. Και πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιοι είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονε που λένε στους ευρωβουλευτές τι τροπολογίε να καταθέσουν. Πολλοί από αυτού είναι ε, τεχνολογικέ επιχειρήσει. Α, ή, ή, ή εκπρόσωποι, ή των ε, οργανώσεων υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως εσύ, Τζο. Ε, προσπαθούμε. Μία από τις εταιρείες αυτές, η eBay, κατέληξε σε μια μελέτη ότι 75% των χρημάτων που δαπανούν οι μεγάλες εταιρείες διαδεθμίσει στο Google χάνονται. Για κάθε ένα δολάριο που δαπανούν, το καθαρό κέρδος ήταν 25 cent. Επιχειρήσεις λοιπόν όπως το Microsoft Πέρσι, νομίζω, δαπάνησε 16,3 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις του Google. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς του eBay, αυτό σημαίνει ότι τα 12 από τα 6 εκατομμύρια ήταν καθαρή ζημιά. Ναι λοιπόν η βιομηχανία έχει απόψεις και πρέπει να την ακούσουμε, αλλά να μείνουν τα πράγματα μέσα σε κάποια όρια. Ευχαριστώ. Αναμένω περιμένω, παραμένω σε αυτά. Κίμον, τι νομίζει, Οι ε, επιχειρήσει λοιπόν παρακολουθούν τη σεξουαλική μας προσανατολισμό. Νομίζω όλοι το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι ο Τζο εν προκειμένου δεν είναι δίκαιος. Εγώ μπορώ να πω και για ομάδες ε, ε θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι πολύ ριζοσπαστικές και κάνουν πολύ ε, ριζικά πράγματα. Το ίδιο ισχύει για την επιχείρηση. Αυτό που ήθελα να πω εγώ προηγουμένω είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπω τα λες. Εγώ δεν γνωρίζω καμιά από τι εταιρείε για τις οποίες εργάζομαι, ούτε ε, διεθνεί, ούτε εθνικές, να μαζεύουν στοιχεία για σεξουαλικέ προτιμήσει. Αυτό που κάνει η διαφήμιση, ο διαφημιστικό τομέα θέλει μεγάλο ε, πεδίο. Κανένας δεν θέλει ένα διαφημιστικό ακόλα σε μένα. Θέλεις να πουλήσεις ένα εκατομμύριο λίτρα αύριο, δέκα εκατομμύρια μπουκάλια παραπάνω αύριο και κάθε μέρα για τα επόμενες τρεις εβδομάδες ας πούμε. Αυτό είναι ο στόχος σου. Άρα χρειάζεσαι ένα μεγάλο τμήμα της κοινή γνώμης. Όσο περισσότερο προχωρήσει να καταλάβει. Αυτά είναι όλα υποθέσεις βέβαια, έτσι. Υπάρχουν, είναι υποθέσεις ότι όταν δηλαδή πηγαίνεις σε μια ιστοσελίδα που είναι για τον γκολφ, σε ενδιαφέρει τον γκολφ. Και πιθανώς 85-90% των περιπτώσεων όντως, αλλά υπάρχουν και 5-10% που ε, έπεσαν κατά τύχη εκεί, το κοίταξαν λίγο, αλλά δεν ενδιαφέρονται για πραγματικά για τον γκολφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, όλα αυτά στη βάση τους είναι υποθέσεις. Όσο περισσότερες λοιπόν υποθέσεις κάνεις, τόσο πιο ακριβές θα είναι το προφίλ του ενδεχόμενου χρήστη που στοχεύει η διαφήμιση της ε, Coca-Cola. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι βασισμένα στα, ε, στα προφίλ είναι πάρα πολύ γενικά ο σεξουαλικό σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μάλιστα και ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, άρα δεν μπορεί κανεί να το επεξεργαστεί χωρίς ρητή συγκατάθεση. Ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλώ. Περίμενα ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων να πει ακριβώς ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται όχι στο profiling. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τη μελέτη του Cambridge. Η ίδια η ιδέα των ευαίσθητων ε, δεδομένων, μήπως σήμερα όλα τα δεδομένα είναι ευαίσθητα. Γιατί με την κατάλληλη τεχνολογία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μεγάλο όγκο πληροφοριών για να καταλήξει και στις ευαίσθητες. Και επαναλαμβάνω και πάλι την ερώτησή μου και σε εσά. Το θέμα της συγκατάθεσης. Μήπως αντί να πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση να μπορεί απλώς να πει ο χρήστης ότι αυτό που κάνω την επόμενε δύο ώρε ή τι επόμενε, ξέρω εγώ, 20 μέρε, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσει κανεί. Απλώ και μόνο. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πάω στην τράπεζά μου και να τους πω όταν θα υπολογίσετε τον κίνδυνο για το ξεπλήρωμα της υποθήκης μου, δεν θέλω να κοιτάξετε αυτό και εκείνο και το άλλο, γιατί τότε θα μου ζητήσετε περισσότερα λεφτά, μεγαλύτερο επιτόκιο, εγώ θέλω χαμηλότερο οι επιχειρήσεις θέλουν περισσότερα συμβόλαια. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ακριβώς γι' αυτό και όχι μόνο για τις δικές μας τις επιχειρήσεις, για όλες τις επιχειρήσεις. Για το θέμα της κατάθεσης όχι, δεν είναι εφικτό. Και μάλιστα θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπατε και εσείς για όλες αυτές τις ε, μικρές πληροφορίες δεξιά και αριστερά που ε, φτιάχνουν, οικοδομούν ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Βάζετε ένα κουκί, ένα κουκί ακριβώς για να μπορείτε να έχετε ε, τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο και η επιχείρηση έτσι μπορεί να ξέρει σε ποιο site πάτε και όχι. Και τι σημαίνει αυτό όλοι αυτοί οι ερευνητές που είναι ακαδημαϊκοί στη θεωρία, στην πραγματικότητα η ζωή είναι τελώς διαφορετική. Θεωρητικά δηλαδή θα μπορούσε κανείς να ξέρει σε ποιο σημείο του website χρησιμοποιήθηκε, πόσο, πότε κτλ. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματική ζωή είναι ότι πας στο ευθύ... εκεί βλέπεις όλες τις κατηγορίες Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ταξινόμηση λοιπόν και ας πούμε ότι έχεις μια κατηγορία FT, Financial Times δηλαδή. Α, άρα αυτός ενδιαφέρεται για τα οικονομικά. Ή πα σε μια ιστοσελίδα για γκολφ και αμέσως βγάζεις το συμπέρασμα αυτός ενδιαφέρεται για τον γκολφ. Και όταν πάτε σε μια άλλη ιστοσελίδα, η επιχείρηση θα δει ότι α, αυτός ε, πάει σε site που είναι και για τον γκολφ και για τα οικονομικά. Δεν πρόκειται για όλα τα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις θέλουν να κρατάνε όσο γίνεται λιγότερα δεδομένα. Άρα τα χρησιμοποιούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό για τη διαφήμιση. Και δεν χρειάζονται όλες τις πληροφορίες. Είναι μύθος ότι οι επιχειρήσεις παίρνουν όλα τα δεδομένα που αφορούν ένα άτομο και τα κρατάνε όλα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν, ξέρουν, δεν θέλουν να ξέρουν τα πάντα για τη ζωή του άλλου. Τα κρατάνε για τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όλα τα δεδομένα λοιπόν δεν ε, συγκεντρώνονται και δεν αποθηκεύονται για καιρό. Ναι, το βασικό όμως, είναι ότι κάποια δεδομένα είναι πιο επικίνδυνα από το καθόλου δεδομένα. Τα μερικά δηλαδή είναι ίσως χειρότερο από το καθόλου μερικές φορές. Και γιατί υπάρχουν αυτά τα κάποια δεδομένα, γιατί κάποιος ε, τα εκμεταλλεύεται και κερδίζει από αυτά. Τον παλιό καλό καιρό που ήταν πιο ακριβή αποθήκευση των δεδομένων, οι επιχειρήσεις ήταν πιο επιλεκτικές στο τι δεδομένα θα αποθηκεύσουν και τι όχι, πάει και έχει περάσει. Τώρα οι καιροί είναι διαφορετικοί. Και κάποιοι, συγκεντρώνοντας ορισμένα από τα δεδομένα σας, μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο κίνδυνο και σε κάποιες φούσκες, για παράδειγμα, που δεν αρέσουν και στους δημοσιογράφους. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει Gmail, η Google αποφασίζει ότι θέλει να ξεκινήσει ένα κοινωνικό δίκτυο, το Google Buzz, και ο κατάλογος επαφών του δημοσιογράφου από το Gmail, εφόσον δεν προβλέπετε τίποτα άλλο, δημοσιεύεται. Ε, δεν ξέρω αν θα σας άρεσε εσάς να γίνει αυτό. Υποθέτω ότι ορισμένοι δεν θα το θέλατε. Η Google λοιπόν δεν θέλει βέβαια να κάνει κατάχραση των ιδιωτικών σας δεδομένων. Από την άλλη μεριά υπάρχει η τάση του να μοιραζόμαστε όσο γίνονται περισσότερα δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα δικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και αυτό είναι που υπογραμμίζω εγώ εδώ. Είναι Είναι Φαντάζεστε ότι από την αρχή της ψηφιακής επανάστασης δεν υπάρχει καθόλου εξέλιξη για το πώς οι επιχειρήσεις ενημερώνουν για την πολιτική του στην προστασία δεδομένων. Το παλιό καλό καιρό με το χαρτί, σας λέω, θα μπορούσα να βάλω ένα χ για να πω ποια δεδομένα θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά και ποια όχι. 17 χρόνια αργότερα από τότε πάσα να ασχολούμαι με το διαδίκτυο, εξακολουθώ να έχω το πρόβλημα ότι η πολιτική για την προστασία δεδομένων είναι χιλιάδες λέξεις και δεν κάθε κανείς να τα διαβάσει. Ακόμα και οι προβουλευτές προσπαθούν να εφεύρουν προγράμματα για να υπάρχει καινοτομία στις επιχειρήσεις, πάση θυσία. Άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Pathfinder do Έχουμε καθόλου επιφυλάξεις ή επιχειρήσεις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ό,τι άλλων για την τοποθέτηση δεδομένων από διάφορες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Είναι μεγάλο το θέμα. Όπως έλεγα και πριν, το να βρει την ε, τοποθεσία όπου βρίσκεται ο χρήστης είναι κάτι που μόλις τώρα αρχίζουμε να εξετάζουμε ακαδημαϊκά. Χρειάζονται ελάχιστα δεδομένα για να βρούμε την ε, τοποθεσία. Αν πάρουμε αυτό που πρότεινε το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Εκείνοι θέλαν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων, να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητε, στα profiling, στις ε, μετακινήσεις, οικονομικές δραστηριότητε, εμπορικές δραστηριότητε κλπ. του ατόμου, που ακόμα και ατομικά ε, οι διάφορες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να έχουν τέτοια πρόσβαση. Άρα λοιπόν πρόκειται για έναν περίεργο κόσμο και είναι ατυχής η στιγμή που έρχεται ο κανονισμός αυτός. Γιατί που πρέπει τώρα, οπότε είμαστε πολύ νωρίς, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς μας συμβαίνει ή περιμένουμε πέντε χρόνια, οπότε τότε θα είναι πολύ αργά για να πάμε πίσω. Και εδώ έχουμε μια ερώτηση, παρακαλώ. Από την Εστονία. Θέλω να ρωτήσω για το profiling. Για το Facebook και την Google, που ως γνωστό φτιάχνουν profiles χρηστών βάσει των πληροφοριών που έχουν από τα ίχνη που αφήνουν οι χρήστες στις διάφορες υπηρεσίες Google ή στο Facebook από τα πράγματα που βάζουν στο τοίχο τους ή τα likes που κάνουν κλπ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα. Γιατί δεν υπάρχει συμφωνία εκ των προπτέρων με το χρήστη ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι ε, εντελώς ανήθικο. Οι στατιστικές που φτιάχνουν οι επιχειρήσεις, οι εφημερίδες που λέγατε που θέλουν να δούνε πόσοι τους διαβάζουν, ποιο άρθρο τους διαβάζουν κλπ. Εντάξει, αλλά η πώληση των προσωπικών αυτών δεδομένων δεν είναι φοβερό. Εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ τη Facebook και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι όχι, δεν πουλάνε προφάιλ. Δεν είναι ότι ο Κίμωνας έχει ένα προφάιλ στο facebook και αυτό πουλάμε. Όχι, αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει το συγκεκριμένο άνθρωπο και προσπαθούν να πουλήσουν στην ε, σελίδα του χρήστη αυτού χώρο για διαφήμιση. Υπάρχουν εκατομμύρια στο facebook οι οποίοι ας πούμε κάποια στιγμή αλλάζουν, λένε ότι παντρεύτηκαν. Οπότε τι συμπέρασμα βγάζουν. Ε, σε κάνα χρόνο μπορεί να έχουν και παιδί. Οπότε μπορεί να αρχίσουν να βάζουν διαφημίσεις για μωρά στην ε, σελίδα facebook του ατόμου αυτού. Αυτό γίνεται. Και μπορείς να πας στο facebook και να δεις πώς γίνεται αυτό. Αυτό αγοράζεις. Το χώρο, το διαφημιστικό χώρο στη σελίδα τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι αυτό που είπα και πριν. Μπορείς να πεις θέλω άντρα ε, στην ηλικιακή αυτή κατάσταση, να βάλεις διάφορες παραμέτρους. Όσο βέβαια πιο λεπτομερής είναι η έρευνά σου, τόσο βέβαια λιγότερα πράγματα θα μπορέσεις να διαφημίσεις άμα είναι πολύ λεπτομερής η έρευνα που έχει κάνει. Άλλες ερωτήσεις για τα λίγα λεπτά που μας μένουν ακόμα. Να, παρακαλώ. Μέχρι τώρα η συζήτηση στράφηκε γύρω από το θέμα πολίτες κατά εταιριών. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που μπορεί να συζητήσουμε αργότερα. Για παράδειγμα αρχές, οργανώσεις κλπ. Όπου πάνε λίγο να φτιάξουν ένα, μια ρύθμιση one size fits all. Για παράδειγμα μπορεί να ισχύει για το facebook αλλά θα έχει και συνέπειες και για πληροφορίες που είναι διαφανείς τώρα για τις αρχές. Και εκεί νομίζω πάμε να μπλέξουμε. Ίσως όμως είναι πρόωρο να θέσω τώρα το ερώτημα. Διερωτώ όμως τόσο αν έχετε κάποιο σχόλιο. Αν εννοείτε τώρα μικρές εταιρείες και πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα. Πρώτα δεν νομίζω ότι είναι θέμα εδώ πολίτες κατά επιχειρήσεων. Είπα πριν ως πρόλογο ότι είναι πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Οι πιο πολλές τροπολογίες που είδα εγώ και είναι και χιλιάδες όλες μαζί δεν πάνε στο συμφέρον της μικρής και μεσαίας επιχείρησης διότι προκαλούν σύγχυση, προκαλούν νομικές δυσκολίες που μπορούν ωστόσο να αντιμετωπίσουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πώς θα περάσει μια μικρή επιχείρηση όλο αυτό τον υπολογισμό δηλαδή βασισμένο ε, στην τεχνολογία, στο ε, επιτόκιο και ούτω καθεξής. Όσο πιο ασαφή είναι τα όρια, όσο πιο θολωμένα είναι τα νερά, τόσο πιο δύσκολο είναι για τι μικρέ και μεσές επιχειρήσεις. Όσο λοιπόν γίνεται αυτό, τόσο μειώνεται η εμπιστοσύνη. Άρα ο κόσμος στρέφεται περισσότερο προς τις επιχειρήσεις τι οποίε εμπιστεύεται. Άρα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ακόμα περισσότερο και την αγορά. Άρα συνολικά εγώ το βλέπω το θέμα ακριβώς αντίθετα από ό,τι το βλέπετε εσείς. Εσείς τώρα. Θα ήθελα να πιστέψω ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μόνο να επεξεργαστούν δεδομένα για να ανοίξουν ε, νέες δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας, κέρδους κλπ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί ξέρω ότι και οι επιχειρήσεις ασκούν και πολιτική. Προσπαθούν να επηρεάσουν τους νομοθέτες, ε, εκλογικές διαδικασίες και άλλα τέτοια και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με την επεξεργασία δεδομένων από τις επιχειρήσεις ότι θα μπορέσουν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους δεδομένα για να ασκήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά επιρροή στις, ε, στην διαμόρφωση ολόκληρων κοινωνιών τι έχετε να απαντήσετε σε αυτού του είδους την ε, βαθιά δυσπιστία. Δεν ξέρω από, από πού προέρχεστε. Εγώ είμαι Έλληνο-Γερμανός. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα τουλάχιστον που είχε ευρύτατα διαδεδομένη δια, διαφθορά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Εγώ μιλώ μόνο για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας και η πολιτική μας δεν λειτουργούν όπως περιέγραψε ο Τζέρεμι, αλλά διαφανώς. Και διαφάνεια για μένα σημαίνει ότι εγώ έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να κάνω την επιχείρησή μου και να ενημερώνω τους πολιτικούς για την επιχείρησή μου. Χτυπάω στην πόρτα τους και αν θέλουν πάω και τους εξηγώ πώς λειτουργεί η αγορά. Γνωρίζω επιχειρήσεις, γνωρίζω τι κάνουν, πώς λειτουργούν στην πλειοψηφία τους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λειτουργούν στις χώρες τους κάτω από την, ε, από την ισχύ του νόμου. Δεν έχω δει ποτέ οτιδήποτε που να προσωμιάζει με αυτά που λέτε. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Αν όμως εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και οι υπόλοιποι εδώ και ο Τζο και οι άλλοι και πάμε στους ίδιους ευρωβουλευτές ε, σε αυτούς που πήγα εγώ ή και θέλω να πάω ακόμη γιατί καμιά φορά οι άλλοι με προλαβαίνουν θα με ακούσουν και θα τους πω την δική μου άποψη. Μα και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι, έχουν κεφάλι και μέσα στο κεφάλι έχουν μυαλό και μπορούν να ακούσουν και να ζυγίσουν τα επιχειρήματα. Το μόνο που λέω εγώ είναι ότι όπως είναι τώρα συνταγμένο το νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και δεν μιλώ εδώ για δουλειές και ανάπτυξη αλλά για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι κυρίως μια υπόθεση business to business και δεν θα δείτε μεγάλες ευρωπαϊκές πλατφόρμες B2C, business to customer, που έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη συγκατάθεση του χρήστη. Ίσως είναι λάθος συζήτηση εδώ για τη συγκατάθεση. Αν ζητήσετε τη συγκατάθεση του χρήστη σε μια μεγάλη πλατφόρμα, ο, ο χρήστης εφόσον το θέλει αυτό που του προσφέρεται θα πει ναι. Δεν θα δώσετε τόσο εύκολα τη συγκατάθεση ωστόσο σε μια εταιρεία B2B, business to business που επεξεργάζεται δεδομένα. Διότι κάνει ένα απλό πράγμα κρατάει τα δεδομένα και διαγράφει τα δεδομένα. Γιατί δεν του χρειάζεται, γι' αυτό δεν θα τι θα δώσει. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι κυρίω B2B. Αν σπρώξετε πολύ το θέμα τη συγκατάθεση, θα πετάξετε λοιπόν αυτέ τι επιχειρήσει έξω από την αγορά. Αυτό θα κάνετε. Και επομένω η business θα πάει στου μεγάλου, στι μεγάλε επιχειρήσει. Αυτό είναι. Δηλαδή η Ευρώπη έρχεται εδώ και νομοθετεί υπέρ τριών, τεσσάρων, πέντε μεγάλων επιχειρήσεων. Τζο. Ναι, φαίνεται όντως να νομοθετεί υπέρ ενός μικρού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν αυτή την προσέγγιση technology based. Είδα ένα τιτίβισμα πριν από λίγο όπου κάποιος έλεγε όταν δίνω τα δεδομένα μου, όταν χρησιμοποιώ ένα κοινωνικό δίκτυο αυτό ε, πάει μαζί με το πακέτο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μου. Αλήθεια είναι αυτό. Αν εγώ ζητήσω ε, έναν ηλεκτρολόγο να έρθει να φτιάξει τα φώτα στο σπίτι μου, ναι, θα έρθει με την προπόθεση ότι θα μπει και μέσα στο διαμέρισμά μου για να τα φτιάξει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει και το δικαίωμα να εγκατασταθεί μέσα στο διαμέρισμά μου και να διαμένει εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εδώ μπροστά. Λέγομαι Stein από την αίση της Γερμανίας. Πού θα βάλετε το όριο ανάμεσα στο κέρδος, στο profit και στο non-profit data. Δεδομένα δηλαδή που συλλέγονται για επιστημονικούς σκοπούς μπορούν μετά να χρησιμοποιηθούν βέβαια για κερδοσκοπικούς λόγους. Νομίζετε ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί κάποια διαφορά ανάμεσα σε, αυτές τις δύο, σε αυτούς τους δύο ε, σκοπούς. Τζο, αν είναι θέμα αξιών κοινωνίας που μπαίνει κάπου στο άρθρο 83, 2 μου φαίνεται, έτσι, κάπου τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο, του κανονισμού, Societal values δηλαδή. Κάτι το οποίο έχει συζητηθεί δηλαδή πρόσφατα. Ναι, μα ποιο αποφασίζει, συνεχίζει ο ερωτών, τι είναι καλό για την κοινωνία. Ποιος βάζει τα όρια. Να ρωτήσετε την ίδια ερώτηση για οποιοδήποτε τμήμα της πρότασης οδηγίας. γιατί μετά καλούν τα δικαστήρια να λάβουν τις αποφάσεις. Δεν μου αρκεί αυτή η απάντηση, διότι τότε απλώς μετατίθεται το πρόβλημα ενώπιον της δικαιοσύνης. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει στη φάση του σχεδιασμού. Ζορμπάς, νομίζω ότι είναι θεμητή ερώτηση, έχετε δίκιο. Και τα άρθρα 82-83 μιλούν για ιατρικά δεδομένα, δεδομένα από έρευνες, Καλά, μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό και επίκριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα τεθεί καν το θέμα, αλλά βασικά μπορεί να, χρησι... τεθεί ένα θέμα, να ληφθούν δηλαδή τα ιατρικά δεδομένα και μετά να φτιαχτεί κάποιο φάρμακο. Ναι, μα τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν συμφωνίες με την βιομηχανία γιατί τα περισσότερα εργαστήρια των πανεπιστημίων χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία. Πού μπορεί να βάλει λοιπόν κανείς εκεί το, το όριο. Ε, εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Πάντα μένει ένα παράθυρο, ένα, ένα δρομάκι ανοιχτό. Και είναι αντιδιοντολογικό αυτό. Κοιτάξτε, τα σχετικά άρθρα όπως είχαν συνταχθεί αρχικά και δεν έχουν αλλάξει και στην προτινόμενη οδηγία, λένε αν χρησιμοποιήσετε δεδομένα για ιστορικούς ε, σκοπούς, ιστορικούς ε, ή επιστημονικούς κλπ, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε δεδομένα ανώνυμα ή ψευδόνυμα. Αυτό έγινε και αντικείμενο κριτική στο προηγούμενο πάνελ. Αλλά παίρνετε τότε τα παρά, τις, παρα, τις παραμέτρους ότι εγώ που έχω κάποιο καρδιακό νόσημα παρόλα αυτά καταναλώνω λίπος αλλά τότε πρέπει να χωριστούν από τις παραμέτρους που ε, επιτρέπουν την ταυτοποίησή μου. Ο ίδιος ο νόμος, δηλαδή, προσπαθεί να αποφύγει ε, το πρόβλημα της πλήρους χρήσης των identifiers, αλλά είναι ένα risk-based approach και επανερχόμαστε στις, ε, στα ψευδόνυμα δεδομένα που είναι βέβαια και γερμανική έννοια και προέρχεται από μια πολύ στενή ε, προσέγγιση που λέει ότι όλα είναι identifiable εκτός αν τα ξεχωρίσετε. Ε, εν τέλει βέβαια είναι υπόθεση των δικαστηρίων όντως. ε, ε, ε η, η κοινωνία των πολιτών δεν καταδικάζει τα ψευδόνυμα δεδομένα Θεωρεί όμως ότι αυτά δεν μπορούν να είναι Όχι, όχι, δεν το, δεν το υποστηρίζουμε αυτό. Υπάρχει συμφωνία στο πάνελ εδώ τουλάχιστον ότι τα ψευδόνυμα δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα. Σχετικό ερώτημα. Το 61F δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να επεξεργάζονται δεδομένα εφόσον θεωρούν ότι αυτό εντάσσεται μέσα στα θεμητά του συμφέροντα. Έχετε δίκιο λοιπόν που λέτε ότι ο, το πεδίο εφαρμογή εδώ είναι πολύ ευρύ. Αλλά χρειά μπροστά στα πεδία που ανοίγει αυτή, αυτή η διάταξη και η Επιτροπή ε, ενιαίας αγοράς εδώ του Κοινοβουλίου είπε ότι ψήφισε μάλλον ότι μπορούν οι εταιρείε να επεξεργάζονται δεδομένα εφόσον τα θεωρούν προς το δικό του συμφέρον και μετά να τα διαβιβάζουν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Και αυτοί οι τρίτοι μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα για σκοπούς που είναι μη συμβατοί με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Να λοιπόν, αν θέλετε παραθυράκι στον νόμο, να παράθυρο και μεγάλο. Υπάρχει πάνελ αύριο στις 11 το οποίο θα ε, συζητήσει ακριβώς αυτά που λέτε τώρα. Είναι πολύ πολιτικό το θέμα αυτό που ε, ρωτάτε και είναι μάλλον θέμα των Ευρωβουλευτών ε, να εξηγήσουν και ποιες είναι οι θέσεις τους. Προτείνω λοιπόν να θέσετε το ερώτημα αυτό αύριο στους Ευρωβουλευτές. Είναι και ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, να πούμε στον τελευταίο γύρο. Okay, so now we're... Καλώς. Μπαίνουμε τώρα στο πιο επίμαχο θέμα. Κατά πόσο ε, μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να μας ξεχάσει το διαδίκτυο. Έχουμε τον Σεμπάστιαν Ντεμπράουρ και την Ούρια Ροντρίκε. Πρώτα ο Σεμπάστιαν Ντεμπράουρ, λοιπόν, που είναι εκτελεστικό διευθυντή τη Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδίας Τραπεζών. Αναφέρθηκε ο τομέα αυτό μέχρι τώρα αρκετές φορές. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, η προστασία των δεδομένων για τις τράπεζες είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι είναι μια συνεχής προσπάθεια που κάνουμε, η προστασία δηλαδή των δεδομένων των πελατών μας και των επενδυτών μας. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε μακριά hackers κλπ μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω τις θέσεις μας για το δικαίωμα να μπορούμε να ξεχαστούμε από το διαδίκτυο. Και ποια είναι η γνώμη μας για τον κανονισμό. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα. Συζητιέται από όλου του ενδιαφερόμενου, από τις χώρε μέλη που λένε ότι θα ζητήσουν εξαίρεση, opt-out για κάτι τέτοιο. Υπάρχει η εποπτεία ε, που, εποπτεία προσωπικών δεδομένων που επίσης εξέφρασε αρνητική γνωμοδότηση. Ίσως βέβαια από την άλλη μεριά εδώ πέρα να δημιουργούνται και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Το νέο άρθρο 17 επιβεβαιώνει ένα δικαίωμα που ήδη υπάρχει, διαγραφής προσωπικών δεδομένων. Κάτι το οποίο αναφερόταν στην οδηγία του 1995. Αλλά το θέμα πάει πιο μακριά. Δεν πρόκειται μόνο για δικαίωμα, διαγραφής εφόσον δεν είναι πλήρη τα δεδομένα ή δεν είναι έγκυρα ή επειδή ο λόγος για τον οποίο ε, τα έχουμε συλλέξει δεν υπάρχει πια. Όχι, υπάρχει και το δικαίωμα του υποκειμένου, του ατόμου, να μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν, εφόσον διαφωνεί με τη διαδικασία επεξεργασίας τους που έχει γίνει. Δεν θα μιλήσω για το δικαίωμα αυτό ευρύτερα, γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι το δικαίωμα αυτό εισήχθη κυρίως για να αντιμετωπιστούν ε, ζητήματα προσφυγής κατά των ε, κοινωνικών ε, δικτύων. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί το δικαίωμα αυτό έχει συνέπειες και στον τραπεζικό τομέα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η πρόσβαση ιστορικά δεδομένα για την ε, οικονομική συμπεριφορά του ατόμου. Στατιστικά έχουν μεγάλη σημασία για τις τράπεζες, για τους δανειστές, γιατί μας βοηθούν να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του ατόμου. Πώς θα αντιδράσει στο δανεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόλις εγκρίνει μια νέα οδηγία για τον υπεύθυνο δανεισμό. Όταν λοιπόν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ένας δανειστής αξιολογεί, ε, τι κάνει, χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει για να καταλήξει σε συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του ατόμου κατά το παρελθόν. Και έτσι αξιολογεί κατά πόσο είναι αξιόπιστος ή όχι ε, αυτός που ζητάει το δάνειο. Όταν ε, λοιπόν ζητάει ένα άτομο τη διαγραφή όλων των προηγούμενων δεδομένων του, τότε οι τράπεζες αλλά και οι πολίτες θα δυσκολευτούν πιο πολύ να καταλήξουν σε συμφωνίες για δάνεια. Γιατί ο δανειστής δεν έχει τίποτα πάνω στο οποίο να μπορεί να βασιστεί για να καταλήξει στο συμπέρασμά του να δανείσει ή όχι τον ετούντα. Αν διατηρηθεί το άρθρο 17, πάντως πιστεύουμε ότι πρέπει, μάλλον ότι δεν πρέπει να επιτρέπει την πλήρη διαγραφή δεδομένων εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι για σκοπό αξιολόγησης, εκτίμησης επιστοληπτικής ικανότητας. Οι οικονομικοί φορείς είναι αλήθεια ότι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους πρόληψης. Για να αντιμετωπιστεί το, η νομοποίηση παράνομου χρήματος οι πάτες Τα δεδομένα δηλαδή που έχουμε από προηγούμενα χρόνια μπορεί κάποια στιγμή να βοηθήσουν να έχουμε το προφίλ του πελάτη. Και εφόσον ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να διαγραφούν τα δεδομένα του αυτό από το παρελθόν, αυτό μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην ε, αποφυγή ε, οικονομικού εγκλήματος. Οπότε το σημείο 17, αν μη τι άλλο, να προσθέσει μία παραπάνω εξαίρεση, που να είναι αυτή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή οικονομικού εγκλήματος, για παράδειγμα. Το κύριο μήνυμα από τη δικιά μας την πλευρά είναι ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές που αναφέρονται στον νέο κανονισμό, κατά τη γνώμη μας, έχουν σχεδιαστεί και διατυπωθεί στα πλαίσια του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων κλπ. Αλλά δεν ταιριάζουν πάντα για την ε, καθημερινή δουλειά των οικονομικών φορέων. Και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η ανησυχία μας πρέπει να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό και θέλουμε να ενημερώσουμε σχετικά τους ευρωβουλευτές. Πιστεύετε ότι πρόκειται όντω για την περίπτωση των τραπεζών μόνο, εδώ πέρα μιλάμε και για κάτι γενικότερο. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ και μπορώ να σας εξηγήσω τι σημαίνει η πρόταση αυτή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι μόνο. Καταρχήν για το δικαίωμα αυτό να ξεχαστεί κανείς από το διαδίκτυο. Ξεχάστε το στο περιβάλλον online το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει. Το δικαίωμα να ζητήσει κανείς διαγραφή των δεδομένων του, λέμε ότι υπάρχει, αλλά υπάρχουν περιορισμοί. Και μερικοί από τους περιορισμούς αυτούς υπάρχουν στην πρόταση. Οπότε συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο απόλυτο δικαίωμα. Υπάρχουν περιορισμοί Ανάλογα με την αναγκαιότητα, αναφερθήκατε και εσείς στον δανεισμό, εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Πολλές φορές στην Ευρώπη υπάρχουν επιχειρήσεις, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σε μερικές, οι οποίες εμπορεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Οπότε γίνεται κατάχρηση. Τα πουλάνε σε τρίτους. Ναι, οι τράπεζες πρέπει να έχουν κάποια δεδομένα στη διάθεσή τους για να ξέρουν σε ποιον πρέπει να δώσουν δάνειο και σε ποιον όχι, αλλά η διαχείριση των μέσων αυτών πρέπει να γίνεται ε, με εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές. Το λέω δεν ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη. Και δεν θα θέλαμε να δούμε στην Ευρώπη περιπτώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων που κρατάνε δεδομένα και τα πουλάνε όπου θέλουν και δεν σας δίνουν το δικαίωμα πρόσβαση σε αυτά, ούτε να τα διορθώσετε και να τα αλλάξετε. Αυτό θα ήταν καταστροφή. Σας παρακαλώ λοιπόν, φροντίστε η διαχείριση των δεδομένων αυτών να γίνεται υπό την εποπτεία των εποπτικών αρχών και να υπάρχουν περιορισμοί για το τι μπορεί κανείς να κάνει και να μην κάνει με τα δεδομένα. Τώρα όταν μιλάμε για το δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς, Πιστεύουμε ότι είναι κάτι θετικό για να προωθήσουμε τον κανονισμό, αλλά από την άλλη μεριά παραπλανεί. Γιατί σας είπα ότι αυτό είναι κάτι ιδεαλιστικό και όχι πραγματικό. Συνεπώς εμείς στηρίζουμε το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και θα υπάρχουν πάντα. Δεν μπορεί δηλαδή να σε ξεχάσει πλήρω το διαδίκτυο. Σήμερα, online, μπορούν να γίνουν παρακλάδια, αντιγραφές των δεδομένων σας που έχετε δώσει στους controllers. Και πολύ συχνά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγραφούν όλα αυτά τα παρακλάδια και, όλες αυτές οι, και όλα αυτά τα αντίγραφα που έχουν γίνει. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή αλλά αυτό έχει να κάνει με τον controller και έχει με τους ενδιάμεσους οι οποίοι πρέπει να είναι ουδέτεροι υπάροχοι δεν είναι και αυτοί οι πάροχοι που μπορούν να έχουν τον περιορισμό. Όχι. Συνεπώς, η προστασία αυτή πρέπει να υπάρξει, πάση θυσία στην αρρύθμιση. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω και μερικά γενικά σχόλια για την πρόταση. Καλή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώς, όπως ακούσατε, πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές υπονόμευσαν και αποδυνάμωσαν πολλές από τις αρχικές διατάξεις. σε σχέση με τον έλεγχο των δεδομένων που μπορούν να κάνουν οι πολίτες. Ένας στόχος του κανονισμού είναι να μπορούν να ανακτήσουν οι πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων τους, κάτι το οποίο το έχουν χάσει. Ο προτινόμενος κανονισμός προσπαθεί να βάλει μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα καλό σύστημα προστασίας από τη μια και από την άλλη να αποφεύγεται οι επιχειρήσεις να επομίζονται η υπερβολικά μεγάλο βάρος. Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες ακούσαμε πολλές παραπλανητικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις που θα έχει πρόταση αυτής της μεγάλες επιχειρήσεις και ξέρετε ποιες είναι αυτές όλοι σας. Δεν είναι αλήθεια όμως, όπως λένε, ότι η, οδηγή, η ρύθμιση αυτή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το διαδίκτυο. Πολλοί λένε ότι θα περιορίσει την καινοτομία μάλιστα. Ε, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ελπίζω πως η πρόταση, αν μη τι άλλο, θα περιορίσει τις παραβιάσεις του νόμου που γίνονται, γιατί πολλές επιχειρήσεις βρουν με τέτοιο τρόπο που παραβιάζουν τον νόμο. Ε, μακάρι αυτό να περιοριστεί. Αλλά για την καινοτομία αυτή καθεαυτή, το αντίθετο από αυτό που είπε ο Τζο θα έλεγα εγώ, ότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη του καταναλωτή, τότε δεν θα υπάρξει καινοτομία. Είναι προϋπόθεση δηλαδή για την ε, καινοτομία να υπάρχει εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ακόμα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΙΜΚΟ ενέκρινε διάφορες τροπολογίες οι οποίες εμποδίζουν ε, τον καταναλωτή να ανακτήσει τον έλεγχο των δεδομένων του. Κάτι το οποίο μας, μας απασχολεί πάρα πολύ και προσπαθούμε σκληρά να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν διάβασα βέβαια και τις 4.000 τροπολογίες, αλλά πολλές από αυτές πάνε σε λάθος κατεύθυνση. Οπότε η πρόταση κανονισμού τι κάνει. Επιβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες αρχές στην τρέχουσα οδηγία. Υπάρχουν δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, το δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα, της διαγραφής τους, της διόρθωσης των δεδομένων, το δικαίωμα ενημέρωσης υπάρχει ήδη. Βέβαια, στο διαδίκτυο, στο online, είναι πιο εύκολο να γίνεται παραβίαση των αρχών αυτών. Οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, οι δυνατότητες ε, Παραβίαση του νόμου που υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο να περιοριστούν. Πολλές επιχειρήσεις παραβιάζουν τον νόμο, μεγάλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα εφαρμόζουν και business models τα οποία δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις και τους νόμους. Έτσι οι καταναλωτές τα έχουν πια χαμένα δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, αλλά η διαφάνεια σημαίνει πολλά πράγματα. Από μόνη τη είναι κάτι θετικό βέβαια, αλλά εξαρτάται πώς την εφαρμόζει κανείς τη διαφάνεια. Συμπέρασμα. Είμαστε στο σκοτάδι για το πώς, γιατί συλλέγονται τα δεδομένα μας, τα επεξεργάζονται κάποιοι και τελικά ορισμένες εταιρείες κάνουν κατάχρηση αυτών. Εννοείται ότι είναι απαράδεκτο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η πρόταση είναι να ανατρέψει την κατάσταση. Η πραγματικότητα και οι πρακτικές δείχνουν ότι η πρόταση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Δεν αναφέρθηκε εδώ, αλλά η Google, μια τόσο γνωστή εταιρεία, έχει μια νέα πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς να έχει προηγουμένως συνανωθεί με τον επόπτη προσωπικών δεδομένων. Και η νέα της αυτή πολιτική παραβιάζει τους νόμους που υπάρχουν και τώρα βρίσκεται βέβαια σε κατάσταση προσφυγής σε βάρος της. Άλλο παράδειγμα, ένα γερμανικό κοινωνικό δίκτυο, το οποίο έκλεισε το 2013, ανακοίνωσε ότι όλα τα δεδομένα και όλο το περιεχόμενο το οποίο είχε συλλέξει και επεξεργαστεί διαγράφεται ανεπιστρεπτή. Ωραία, προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό. Τέλος, πολλές επιχειρήσεις που σας πουλάνε στο ίντερνετ και όχι μόνο στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και τους δίνετε την πιστοτική σας κάρτα, τον αριθμό της πιστοτικής σας κάρτας τον κρατάνε και τον χρησιμοποιούν για άλλους λόγους από τους οποίους εσείς τους δώσατε τα δεδομένα αυτά. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική, τι καταχρήσεις γίνονται και τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αυτές. Κάποια στατιστικά δεδομένα Τώρα που λένε ότι οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα, και αυτό συμβαίνει παντού, ε, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν οι ευρωβουλευτές να μην ακούν ότι το 70% των καταναλωτών λένε ότι τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους από αυτούς για τους οποίους τα έχουν δώσει σε εταιρείε. Λένε επίση ότι 67% δεν έχουν εναλλακτική λύση αν θέλουν να αγοράσουν κάτι, κάποια υπηρεσία, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν την πιστοτική τους κάρτα. Δηλαδή, μερικές φορές ή που δίνεις την πιστοτική σου κάρτα, τα προσωπικά σου δεδομένα, ποια και αν είναι αυτά, ή αλλιώς δεν έχεις την υπηρεσία που θέλεις. Το βροβαρόμετρο δε λέει ότι ακριβώς η έλλειψη αυτή εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι εκείνη η οποία εμποδίζει την ε, καινοτομία και την ε, ανάπτυξη του εμπορίου. Άρα, αποτελούν πλεονέκτημα και όχι βάρος. Έτσι θα έπρεπε να το βλέπουν και οι επιχειρήσεις. Γιατί το κέρδος αυτό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αν ο καταναλωτής είναι ενημερωμένο. νιώθει ότι υπάρχει διαφάνεια και έχει εμπιστοσύνη, με μεγαλύτερη άνεση θα αποφασίσει να δώσει και τα δεδομένα του. Θέλω να πω δύο λόγια τώρα για ένα νέο δικαίωμα. Αντίθετα με αυτό για το να ξεχαστεί κανείς από το δίκτυο, που δεν λέω ότι διαφωνούμε με την ιδέα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ισχύει καλά, είναι το δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων. γιατί και αυτό έχει να κάνει με το δικαίωμα πρόσβασης ή με το δικαίωμα ελέγχου του τι γίνεται με τα δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο δίκαιο το οποίο μπορεί να κάνει τους καταναλωτές να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιείται ένα κοινωνικό δίκτυο ή μια πλατφόρμα που αποθηκεύεται τις φωτογραφίες σας και διαπιστώνετε ότι ο σερβερ σας έχει εξαπατήσει, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να σβήσετε την επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει μέχρι τώρα, έχει συμβεί μερικέ φορές και δρά θετικά στον ανταγωνισμό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτό στο μελλοντικό κανονισμό, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε ερωτήσεις. Εσείς. Από την Εσθονία. Και επανέρχομαι στην κυρία Ροντρίγκεζ. Από αυτά που κατάλαβα, από αυτά που είπατε, ότι οι εταιρείε είναι κακές, δεν μπορεί να σε εμπιστεύεται κανένας και κάθε τι που κάνουν με τα δεδομένα θα πρέπει να αστυνομεύεται από τις αρχές. Ναι, αλλά ποιος θα το κάνει αυτό και ποιος θα το πληρώσει. Θα μας προσλάβουν οι κυβερνήσεις όλους μας για να αστυνομεύουμε τα δεδομένα. Απάντηση. Δεν είναι απόλυτα σωστό. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα ότι πρέπει να αστυνομεύεται από τις αρχές και μάλιστα το κάθε τι. Η πρόταση νόμου με την κατάργηση της υποχρέωσης κοινοποίησης διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Ένα από τα προβλήματα Τη συμμόρφωση με τις ε, αρχές προστασίας των δεδομένων είναι ότι οι κανόνες δεν επιβάλλονται. Η πρόταση που συζητούμε προβλέπει ένα αριθμό διατάξεων που θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής να επιβάλλουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις αρχές προστασίας των καταναλωτών. Άρα, όντως χρειάζονται πόροι για αυτό, συμφωνώ αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης και μια καλή οργάνωση. Ότι δηλαδή οι αρχές προστασίας των δεδομένων είναι καλά οργανωμένες και ότι δι γίνεται επικάλυψη έργου και επομένως απώλεια χρόνου. Και νομίζω ότι η κατεύθυνση της πρότασης εδώ είναι ορθή. Δηλαδή οι αρχές επιβολής του νόμου να εργάζονται αποτελεσματικά. Βέβαια θα χρειαστούν περισσότερους πόρους, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Άλλος κανείς, άλλη καμία. Εγώ να συνεχίσω από τη δική σας ερώτηση. ερώτηση. Μιλήσατε για την υπόθεση του Google και πώς επέκτηναν την privacy policy και με ένα αριθμό παραπώνων. Αναμένουμε ακόμα αποφάσεις. Γιατί νομίζετε ότι ακόμα αναμένουμε τις αποφάσεις. Τι να σας πω, πράγματι η ερώτηση ε, για να σας απαντήσω είναι ατυχές. Ελπίζαμε οι αρχές προστασίας των δεδομένων, ελπίζαμε, ελπίζαμε ότι η Google θα συμπεριφερθεί σωστά και πριν να αρχίσει να εφαρμόζει νέα πολιτική θα προχωρήσει σε πλήρης διαβουλεύσεις με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Αυτό το πρώτο πράγμα που ελπίζαμε και βέβαια πρέπει να ζητήσουμε και από τις αρχές προστασία των δεδομένων να δράσουν ταχύτατα. Εκτός αν αποφασίσετε όλοι ότι δεν θα χρησιμοποιείτε πλέον το Google, αλλά από ό,τι βλέπω όλοι το χρησιμοποιείτε. Εσείς όχι για το θέμα αυτό, εκτός ίσως από ένα σχόλιο συμφωνούμε σε πολλά από τα θέματα με την κυρία Ροντρίγκε. Για παράδειγμα για τα δεδομένα για την πιστοληπτική ικανότητα. Χρειάζονται βέβαια κάποιες εξαιρέσεις. Με το πρώτο σχέδιο δεν ήταν αρκετές οι εξαιρέσεις αυτές. Αυτές ήδη εν μέρη διορθώθηκαν. Είπατε η ίδια ότι πολλές επιχειρήσεις δεν σέβονται ή δεν συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει αυτό με τη νέα νομοθεσία. Αυτό που είναι σημαντικό νομίζω στα όσα είπατε είναι η ανάγκη της επιβολής. Πρώτα να συμμορφωθούν οι εταιρείε με την νομοθεσία του 1995 και αυτή είναι εφαρμοστή, είναι πρώτη προτεραιότητα, έτσι θα Ναι, είναι πολύ σημαντικό, λέει η κυρία Ροντρίγκε, να φροντίσουμε ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρώσεις τους. Υπάρχουν πολλές παλαιές ας πούμε αρχές στην πρόταση που δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικές, είναι πολύ σημαντικές. Και νέες ε, διατάξεις που επιβάλλουν συμμόρφωση της βιομηχανίας με, την, ε, με τις ε, αρχές αυτές. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι η επιβολή είναι σημαντική και είναι και από τα κύρια προβλήματα. Βέβαια πρέπει να πει κανείς ακόμη ότι αντιμετωπίζουμε, με ένα, αντιμετωπίζουμε ένα περιβάλλον online όπου βέβαια είναι σαφές ότι είναι πολύ ευκολότερο να παραβιαστεί ο νόμος στον εικονικό κόσμο, στον virtual κόσμο από ότι στον πραγματικό. Οι επιχειρήσεις λοιπόν χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται την ευκαιρία αυτή που έχουν. Που έχουν. Και βέβαια πάντα ο νόμος τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Στην πραγματικότητα όμως νομίζω ότι είναι σωστό το χρονικό σημείο και πρέπει τώρα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς θα γίνει ακόμα χειρότερο στο μέλλον. Είναι λοιπόν κάπως αργά βεβαίω, αλλά δεν είναι ας πούμε πολύ αργά. Θα πρέπει να έχουν και άλλες ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Εσείς. Σουηδία. Πριν από ένα χρόνο και περισσότερο, μια έκθεση δημοσιεύτηκε από το European Network για την ε, ε, ασφάλεια των δεδομένων στο διαδίκτυο και νομίζω ότι είναι μια αρχή που είναι κατεστημένη στην Κρήτη και είχαν πει ότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτή, αυτό σε ανοιχτά δίκτυα. Αυτή η έκθεση βρήκε κάποια απήχηση στη συζήτηση ή μιλούμε για κάτι το οποίο είναι απολύτως υποθετικό. Νομίζω ότι η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά έχετε δίκιο. Η έκθεση είναι σημαντική και αυτά που είπα αρχικά στη συζήτηση, παρόλο που κυρίως αναφέρονται στο τραπεζικό τομέα, δέχτηκα ωστόσο ότι αυτή η συζήτηση προκαλεί και εσφαλμένες προσδοκίες, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι ευρωβουλευτές βέβαια που εξακολουθούν να συζητούν το θέμα αυτό, πιστεύω θα συνεχίσουν να το συζητούν. Εσείς με το λευκό υποκάμισο. Ναι, από την Τσεχία. Εσείς ταχθήκατε υπέρ της συλλογής των δεδομένων με υπεύθυνο τρόπο κλπ. Αλλά οι αρχές συλλέγουν πολλά δεδομένα. Όχι μόνο για ποσά χρημάτων που δανείζουν ή δανείζονται οι ορισμένοι, αλλά και πληροφορίες και για πιστοτικές κάρτες και άλλα σχετικά εργαλεία, που βεβαίως αυτά είναι πηγή πολύτιμων πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ε, κρατικές αρχές αλλά και άλλες επιχειρήσεις Ούτε είναι ωραίο αυτό για, το, για τους πολίτες να είναι κάτω από τέτοια πίεση των τραπεζών που αυτές μπορούν να παρακολουθούν τι ακριβώς αγοράζουν ή πολλούν ή οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα. Δεν μπορεί να είναι απεριόριστη η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων γιατί αυτό γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο για τους απλούς ανθρώπους. Μπορεί να είναι ωραίο για τις τράπεζες, μεγάλες ή μικρές αλλά όχι για τον κόσμο. Τι λένε οι Δεν ε, εκπροσωπώ τις αρχέ που μιλήσατε, που, που αναφέρατε, αλλά όντως συλλέγονται δεδομένα στις τράπεζες. Δεν γνωρίζω ωστόσο τράπεζες που κάνουν προφίλ των πελατών τους στη βάση πληρωμών προς καταστήματα. Δεν νομίζω να ενδιαφέρονται οι τράπεζες για τέτοια πράγματα. Βέβαια θα έχουν τα δεδομένα των ε, πράξεων που κάνετε εσεί μέσω των τραπεζών τους. Αυτό βέβαια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ακραία τα πράγματα, ξαναλέω. οι τράπεζες θα πράξουν πάντο δυνατό για να κρατήσουν τα δεδομένα για τους εαυτούς τους. Καμιά φορά μας κατηγορούν μάλιστα ότι είμαστε υπερβολικά προστατευτικοί για τα δεδομένα των πελατών μας. Αυτό όμως είναι, έχει μεγάλη, αυτά έχουν μεγάλη αξία. Είναι high value για τις τράπεζες. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε, λέει κ. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω σχετικά με την χρήση που επιφυλάσσουν στα δεδομένα αυτά οι τράπεζες που έχουν συλλέξει δηλαδή για τον αποκλειστικό σκοπό ε, να δανείζουν δηλαδή με υπεύθυνο τρόπο. Ένα θέμα που μας ανησυχεί είναι ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή να αποφασίσει κάποια τράπεζα αν έχει το δικαίωμα να ανοίξετε το τραπεζικό λογαριασμό ή όχι, γιατί εκεί δίθεται θέμα financial inclusion, να μην αποκλείεται κανένας δηλαδή από το να έχει τραπεζικό λογαριασμό κτλ. Δεν έχω βαθιά γνώση το τι κάνουν οι τράπεζες, τι κάνει η τράπεζά μου με τα, δεδομένα μου. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να σχολιάσω περισσότερο. Και εκεί κάπου μια ερώτηση, κάπου, δηλαδή ήταν τρία χέρια πριν, δύο μιλήσανε. Αλλά τώρα το τρίτο χέρι χάθηκε. Ίσως να πούμε και κάτι για, το, για τη φιλοσοφική πτυχή των δεδομένων ή των δικαιωμάτων, κάτι που απασχολεί τους νόμομαθείς όσο περιμένουμε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίσει για το δικαίωμα να λησμονηθεί κανείς. Ορισμένοι από εμάς γνωρίζουμε την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου που κάποιος καθυστερούσε τις πληρωμές για το δάνειο για το σπίτι του και ζητεί τώρα να διαγραφούν όλα τα σχετικά δεδομένα από το Google και από άλλα. Υπάρχει και άλλη μια υπόθεση στις Ενωμένες Πολιτείες, κάποιος δηλαδή που είχε παραβεί τον νόμο για τα ναρκωτικά, μια γυναίκα μάλιστα, και διαγράφηκε η καταδίκη της. Και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διαγραφούν τα σχετικά δεδομένα μιας καταδίκης δηλαδή, στη, από το διαδίκτυο κτλ. Και αυτή η υπόθεση ήρθε ενώπιον των δικαστηριών στο Connecticut. Αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να βρει δουλειά, διότι στο Google βρίσκανε οι, πιθανοί, οι ενδεχόμενοι εργοδότες τα σχετικά με την καταδίκη της. Λοιπόν, αυτό τι είναι, είναι δίκιο Δύσκολη φιλοσοφική ερώτηση απαντούν οι τράπεζες. Εδώ μπαίνουν δύο θέματα. Αφενός νομίζω πρέπει να γίνει μια διάκριση στην, ε, από τη μια μεριά δηλαδή στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και από την άλλη μεριά στη χρήση τους. Και στην περίπτωση αυτή η διάκριση, ίσως και ανεπίτρεπτη χρήση των δεδομένων. Εδώ αυτά νομίζω είναι ξεχωριστά πράγματα. Δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα από τον τραπεζικό τομέα. Για παράδειγμα μιας ποινική καταδίκης στο παρελθόν που δείχνει ότι για παράδειγμα δεν επιστρέψατε ένα ποσό είναι όμως αυτή ε, χρήσιμη προφορία για το αν θα πάρετε άλλο δάνειο. Αυτό όμως δεν μπορεί να σας ε, να αποτρέψει από το να σας προσλάβουν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή άλλο είναι να, μην μπορείτε να βρείτε δουλειά για το λόγο αυτό. Επομένως, τίθεται και το θέμα του σκοπού για, του, για τον οποίο συλλέχθηκε το δεδομένο. Εδώ νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανεί ότι ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους, one size fits all. Το θέμα τώρα για το δικαίωμα να λησμονηθεί κανείς ή τα όρια του δικαιώματος αυτού, το δικαιώματο τέλο πάντων της διαγραφής των δεδομένων σας. Ναι, εδώ βέβαια πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία. Υπάρχει και η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της αναζήτησης πληροφοριών. Εξαρτάται από την περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπερισχύσει το ένα δικαίωμα, σε άλλη περίπτωση θα υπερισχύσει το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και ούτω καθεξής. Επομένως, θα έλεγα, ας αφήσουμε καλύτερα τους δικαστές να κρίνουν. Ε, άλλες ερωτήσεις εκεί πίσω η κυρία. Είμαι Ελληνίδα δημοσιογράφος, όπου και συνάδελφοι που, ο συνάδελφος μου μίλησε πριν. Έχω μια ερώτηση, γιατί κάτι ε, έχει συζητηθεί πολύ και θα ήθελα να ακούσω κυρίως από την κυρία Ροντρίγκες, που ε, προέσταται οργάνωσης καταναλωτών. Ποιος κληρονομεί τα δικαιώματα επί των δεδομένων. Αυτό βέβαια το ερώτημα πάει και στους δυο σας. Δεν έχω διαβάσει όλες τις τροπολογίες επί της οδηγίας. Δεν είμαι βέβαια ωστόσο ότι το θέμα αυτό έχει διευκρινιστεί. Κάποιο λοιπόν χορηγεί τα δεδομένα του, δίνει και την συγκατάθεσή του, όμως όταν πεθάνει το πρόσωπο ή δεν είναι πλέον ικανό να χειρίζεται τα δεδομένα του, τι είδου νομοθεσία εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση, μετά δηλαδή. Ή για παράδειγμα δεδομένα παιδιών. Δεν το έχουμε δουλέψει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Η πρόταση της Κομισιόν ούτε και αυτή το λύνει το πρόβλημα. Δεν έχει κανένα ειδικό άρθρο γι' αυτό. Τώρα, λογικά επιχειρηματολογώντας θα έλεγα ότι το κληρονομικό δίκαιο πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά τι να σας πω, δεν το ξέρω κιόλα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά Facebook, Google και τέτοια πράγματα, αυτά τα δίκτυα δηλαδή, δεν εφαρμόζουν το κληρονομικό δίκαιο. Υπάρχει μέγα πρόβλημα εδώ και διεθνώς. Νομίζω ότι όντω εφαρμόζεται το αστικό δίκαιο, λέει ο κ. Ζορμπά, το θεμελιώδε πρόβλημα που βλέπω εγώ στην πρόταση τη Κομισιόν. Αν και στην ουσία του δεν μα προκαλεί μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι η Κομισιόν είναι ότι πάει να χώσει ό,τι μπορεί μέσα στην πρόταση αυτή. Data portability, μικρό μέγα θέμα, είναι άλλο. Δεν έχει σχέση με προστασία δεδομένων. Δεν πρόκειται για δεδομένα δεν μπορείτε να επεκτείνετε την προστασία δεδομένων, να καλύψει τα πάντα που έχουν σχέση με τα δεδομένα σας. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι σωστότερη ε, πτυχή του δικαίου που θα πρέπει να εφαρμοστεί από το να δημιουργηθεί ένα νέο δικαίωμα προστασίας δεδομένου. Αστικό δίκαιο εδώ. Ορισμένες επιχειρήσεις το δέχονται, άλλες όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχει και μια βραζιλιάνικη υπόθεση που έχει ε, αποτελέσει αντικείμενο ενός τιτιβίσματος και το δικαστήριο εφάρμοσε βραζιλιάνικο δίκαιο. Ούτε θυμάμαι ποια, ποια μεγάλη αμερικανική εταιρεία και ε, διέταξε το δικαστήριο να κλείσουν μια σελίδα προφίλ. Άλλο θέμα της δικαιοδοσίας. Επίσης πολύ προβληματικό. το δικαίωμα στο data portability που λέτε ότι δεν είναι θέμα ε, προστασίας δεδομένων. Εγώ δεν συμφωνώ. Τα προσωπικά δεδομένα που μεταβάζονται, που τα δίνουμε κάπου και τα επεξεργάζονται οι άλλοι, εξακολουθούν να είναι δικά μας δεδομένα. Το δικαίωμα πρόσβασης πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Ελπίζω να συμφωνείτε το δικαίωμα στο data portability είναι ένας άλλος τρόπος για να μπορούμε να ζητήσουμε έλεγχο ή να ανακτήσουμε τα δεδομένα μας. Ακόμα και αν δεν κολλάει καλά στον κανονισμό, πρέπει να ισχύει, γιατί αλλιώ υπάρχει μονοπόλιο. Ακόμα και αν ορισμένοι νομίζουν ότι δεν έχει άμεση σχέση με την προστασία δεδομένων. Μα το είπατε ότι είναι θέμα ανταγωνισμού. Σωστά. Άπαξ και μία ε, επιχείρηση κυριαρχή. Ναι, αλλά ακριβώ οι καταναλωτέ είναι εκείνοι οι οποίοι με τη συμπεριφορά του θα οδηγήσουν στην ε, ανταγωνιστική αγορά. Παλιά ήταν κάτι διαφορετικό ανταγωνισμό από τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ τώρα υπάρχει πλήρη σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Συμφωνώ για αυτά που λέτε για τον ανταγωνισμό. Το στοιχείο κλειδί πάντως είναι ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ή να τα μεταφέρει, αλλά αυτό πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα τα οποία εσείς προσωπικά έχετε παραχωρήσει. Γιατί αυτή ήταν η πρώτη ιδέα στην πρώτη πρόταση. Για το κατά πόσο πρόκειται για δεδομένα που έχουν κάποιοι άλλοι επεξεργαστεί και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους. Και αυτό πάει πολύ μακριά. Συμφωνώ ότι χρειάζεται διευκρίνηση πάντως. Ωραία. Άλλη ερώτηση εκεί πίσω για το δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς στο διαδίκτυο. Είμαι και εγώ δημοσιογράφος από την Ελλάδα και θέλω να ρωτήσω για το δικαίωμα αυτό. Αν δώσω τη συγκατάθεσή μου για να διαγραφούν τα δεδομένα μου, Το δικαίωμα αυτό όμως αναδημοσιεύεται από άλλες ιστοσελίδες. Οπότε ρωτάω, η ιστοσελίδα πρέπει να ανοιχνεύσει ποια άλλα, ποιες άλλες ιστοσελίδες έχουν αναδημοσιεύσει τα δεδομένα μου ή είναι ο κοντρόλερ που το κάνει αυτό. Την υποχρέωση κανονικά την έχει ο κοντρόλερ. Εκείνος πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα που έχουν τύχει επεξεργασία. Αλλιώ δεν θα γινόταν. Όσον αφορά τώρα για του πάροχου, host providers, το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι ότι η οδηγία όταν φτιάχθηκε το 1995 δεν είχε στο νου τη, το διαδίκτυο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι δικαστές είναι αντιμέτωποι με όλη τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Προς το παρόν είναι δύσκολο πάντως αυτό το θέμα. Η ουσία του θέματος, του θέματος γιατί είπαμε στην αρχή ότι δεν είναι ρεαλιστικό να ξεχαστεί κανείς πλήρως από το διαδίκτυο, είναι γιατί το βάρος είναι τεράστιο που πέφτει στους κοντρόλες. Πρώτα απ' όλα πώς να ελέγξει την ε, χρήση των δεδομένων αυτών εφόσον αναδημοσιεύονται σε άλλες ιστοσελίδες. Οπότε κατά πόσο κάποια μέρα θα είναι ρεαλιστικό το να μπορούμε να ξεχαστούμε πλήρως, δεν ξέρω. Άλλες καυτές ερωτήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω το πάνελ μου πως υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που έχουμε ξεχάσει. Εσείς, ας πούμε, από τη ζωή σας, έχετε κάποια δεδομένα που θα θέλατε να ξεχαστούν πλήρως. Όχι. Εγώ χρησιμοποιώ κάτι άλλο, όχι τον Google, που δεν ε, συλλέγει δεδομένα. Και έτσι προσπαθώ να προστατεύω τον εαυτό μου μέχρι να αποσαφανιστεί η κατάσταση. Ε, προσπαθώ, πώς προστατεύω τον ιδιωτικό μου βίο βασικά, αυτό ρωτάτε. Τα email σας, εσείς ξέρετε που αποθηκεύονται. Καμία ιδέα. Εγώ την τάση να πω όχι, δεν, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Να ρωτήσουμε τη Microsoft. Ωραία. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να τις απευθύνετε και στον ε, επόπτη προσωπικό δεδομένο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη, Κλέρ. Μια στιγμή από πλευρά της οργάνωσης. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που συμμετείχατε στο πάνελ αυτό, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, Και τώρα, αν έχετε χρόνο και θέλετε, ελάτε στον πέμπτο για ένα ποτό. Όπως είπε και η Κλέρ, αύριο θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις ερωτήσεις σας στους Ευρωβουλευτές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.